Καλημέρα συνάδελφοι. Herzlich Και καλώ ήρθατε στη συνεδρίαση τη Επιτροπή μα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα για τη σημερινή ημέρα και αύριο το πρωί με ένα μαραθώνιο ψηφοφοριών. Να υπενθυμίσω σε όλους να φέρουν τις κάρτες ψηφοφορίας αύριο το πρωί. Dann beginnen wir heute mit unserer Tagesordnung, die sich να ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Έχουμε δύο αλλαγέ στο σημείο παριθμών 9 για τις ε, διαδικασίες ε, δραστηριότητες της ΣΤΟΑ. Αναβάλλει το θέμα αυτό για κάποια άλλη συνεδρίαση. Και για το θέμα για την φαρμακο... φαρμακοεπαρή το 19. Θα το αναβάλουμε για την επόμενη συνεδρίαση. Το ζήτησε η συγγήτρια. Έχετε άλλα σχόλια για την ημερήσια διάταξη. Αν όχι, εγκρίνεται λοιπόν ως έχει. Wir haben ein TV bei uns, und zwar unser eigenes von äh, DG IPOL, die äh, einige Szenen aus dem Umweltausschuss έχουμε μαζί μας ε, κάμερες. Να σας ε, προειδοποιήσω ότι αύριο θα έχουμε πιο πολύ κόσμο. Μην δώσουμε και λάθος εντυπώσεις. Θα έχουμε πιο πολύ κόσμο αύριο. Νούμερο 2. Στο 2. Στις ανακοινώσεις να σας πω ότι αύριο δεν θα έχουμε μαλτέζικα. Επίσης να αναφέρω ότι ο Μπανκιμούν, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, έδωσε εντολή στο Academy Council στην Ολλανδία να ελέγξει τα, την εργασία, το έργο της IPCC. Αυτό το καλωσόρισε η πλειονότητα και εγώ χαιρέτησε το γεγονός ότι δίνεται τέτοια εντολή σε ένα επιστημονικό σε μια επιστημονική οργάνωση, όχι σε μια κυβερνητική διοικητική οργάνωση, γιατί νομίζω ότι η επιστήμη του κλίματος θα πρέπει να είναι ουδέτερη και ανεξάρτητη και το, αυτό το Academy Council είναι ένα επιστημονικό ίδρυμα το οποίο χαίρει υψηλού κύρους και ελπίζουμε να προσδώσει νέο κύρος στο έργο της IPCC, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξέδωσε μία ανακοίνωση για τη βιώσιμη δασοκομεία, ενδιαφέρον θέμα αυτό, μας ενδιαφέρει και εμάς. Θα ασχοληθούμε με αυτό και θα ασχοληθούμε με αυτό στο μέλλον. Να περάσω στο 3 τώρα στην μερίσια διάταξη. Η οδηγία για την ξυλία. Το Συμβούλιο την 1η Μαρτίου εξέδωσε την ε, κοινή του θέση. Και έτσι μπορούμε να περάσουμε στη δεύτερη ανάγνωση. Στο σημείο λοιπόν αυτό έχουμε μόνο το χρονοδιάγραμμα στη διάθεσή μας. Να σας το ανακοινώσω. Το σχέδιο σύστασης της ε, Caroline Λούκας θα το ψηφίσουμε στις 7 Απριλίου. Θα το εξετάσουμε μάλλον στις 7 Απριλίου. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών 8 Απριλίου, μικρό, μικρή προθεσμία. 3-4 Μαΐου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια του Ιουλίου επίσης θα περάσει το θέμα αυτό. Να προχωρήσουμε λοιπόν στο 4 της ημερήσιας διάταξης. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής θάλασσας και ο ρόλος των μακροπεριφερειών στην μελλοντική πολιτική συνοχής. Η εισηγήτρια, η κυρία Άννα Ρόσμπαχ, θα μας κάνει μια εισαγωγή στην έκθεση. Έχετε το λόγο. Ja, det er jo Ευχαριστώ. Έχουμε μια ιστορία από την Επιτροπή Περιφερειών σε ό,τι αφορά την περιοχή της Βαλτικής θάλασσας και την σχετική στρατηγική και έχω εδώ τονίσει τα θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής στην, ε, στο έγγραφο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν έχει υπογραμμιστεί ιδιαίτερα αυτή η περιβαλλοντική πτυχή. Εδώ μιλάμε λοιπόν για τις μακροπεριφέρειες και φυσικά είναι φυσιολογικό το γεγονός ότι ασχολείται η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης με αυτό το θέμα, γιατί όμως θεωρούμε ότι θα πρέπει να περιληφθούν και άλλα στοιχεία για τη Βαλτική. Δεν είναι μόνο η θάλασσα περιλαμβάνονται και οι όμορες χώρες και φυσικά αυτό άπτονται και θεμάτων περιβάλλοντος. Προσπαθούμε λοιπόν ε, να αναφερθούν και περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η απόρριψη επικίνδυνων ουσιών. Και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία αποτελούν τμήμα του όλου προβλήματος, γιατί ε, περνάει και ο στόλος τους από εκεί. Καλούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη και τα περιβαλλοντικά αυτά στοιχεία. Ασχολήθηκα λοιπόν και με θέματα και συζήτησα και με άτομα που ασχολούνται με το North Stream. Δεν είναι ενθουσιασμένοι. Ελπίζω να μάθουμε πιο πολλά στοιχεία και στη διάρκεια της σημερινής ημέρας για το θέμα αυτό. Είναι κρίμα που δεν λαμβάνονται υπόψη όλα τα συμπεράσματα. Πρόκειται για κάτι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Και η στρατηγική αυτή, αν θέλετε, αποτελεί μια συνέχεια, μια αντίστοιχη πολιτική σε ό,τι αφορά τη στρατηγική για τη Μεσόγειο και για άλλες θάλασσες. Ε, αν μόνο λοιπόν να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων, δεν ξέρω αν θέλει κάποιο να κάνει και προσθήκες. Όπως και να έχει, θα χαρώ να λάβω σχόλιά σας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν υπάρχουν παρατηρήσει. Εγώ να κάνω, αν μου επιτρέπετε, μία μικρή παρατήρηση. Η κυρία Ρόσπαχ ανέφερε τον Äh, Φυσικά πρόκειται για μια παρέμβαση στην ε, Βαλτική θάλασσα, αλλά το γεγονός αυτό που αναφέρεται στο σημείο 4 ότι το Nord Stream θα έχει μεγάλο αντίκτυπο για την περιοχή, ίσως να προκαταβάλει υπερβολικά αν θέλετε τα πράγματα, γιατί Τέσσερα κράτη άλλωστε έχουν ελέγξει το Nord Stream, η Φιλανδία, η Σουηδία, η Λιθουανία, αν δεν κάνω λάθος, και η Γερμανία έχουν ελέγξει αυτό το project, το έργο αυτό. Τώρα αναφέρεται μακροπρόθεσμες και εκτεταμένες ε, επιπτώσεις ότι θα έχει το project αυτό. Δεν είμαι βέβαιος, μήπως ε, υπερβάλλουμε λίγο. ότι μπορεί να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, το δέχομαι, αλλά ότι θα έχει μακροπρόθεσμες και εκδομένες ε, επιδράσεις δεν ξέρω. Ο Ρίχτατ Σέιμπερ. Πρόεδρε, δεν ξέρω αν κάνετε τις παρατηρήσεις ε, που κάνατε ως ε, μέλος ή ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή η έκθεση της κυρίας Ρόσμπαχ. Και εγώ έχω τις αμφιβολίες μου σε ό,τι αφορά τον αγωγό αερίου Nord Stream. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι η συγγήτρια ακολούθησε σωστή προσέγγιση και έβαλε αν θέλετε στο επίκεντρο τα θέματα τα περιβαλλοντικά στην έκθεσή της. Συνολικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να τονίσουμε ίσως λίγο παραπάνω το θέμα των μακροπεριφερειών και να δώσουμε και λίγο παραπάνω περιεχόμενο. Όπως ξέρετε γίνεται και στην Επιτροπή εμ, Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, σχετική, σχετική συζήτηση και ίσως θα έπρεπε από δική μας πλευρά, από πλευρά της Επιτροπής Περιβάλλοντος, να δώσουμε και εμείς λίγο ε, παραπάνω περιεχόμενο. Για παράδειγμα, τη στρατηγική για την ε, γενικότερη περιοχή να σκεφτούμε μήπως θα πρέπει να τεθούν και περιβαλλοντικά ζητήματα. Να μην δηλαδή απομονωθούν μόνο κάποια θέματα για τη Βαλτική θάλασσα, να δοθεί ένα γενικό πλαίσιο Αλλά από την άλλη να πω ότι μου αρέσει η προσέγγιση γενικά της συγγήτριας και την ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Μαρίτα Ουσκόκ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω σου ειδικά. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της. Πραγματικά έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταρτήσει μια σωστή πολιτική για τη Βαλτική θάλασσα που θα περιλαμβάνει και συγκεκριμένες πτυχές ε, για το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να κάνουμε και ό,τι μπορούμε για να πραγματοποιήσουμε τη στρατηγική αυτή. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε δηλαδή στα ωραία λόγια, στις ωραίες δηλώσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν και πραγματικότητα, γιατί εκεί είναι το πραγματικό πρόβλημα, το ουσιαστικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη Βαλτική θάλασσα τώρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι τα μέτρα που έχουν ε, ληφθεί θα πρέπει να εκτελεστούν, να εφαρμοστούν, να πραγματοποιηθούν. Και αυτό δεν έχει γίνει έως τώρα. Όλες οι προτάσεις έχουν μείνει στο κενό. Καλό λοιπόν θα ήταν αυτό κάπου να καθίσταται σαφές και στο κείμενο. Κάπου στην έκθεση δηλαδή να πούμε με σαφήνεια ότι είναι σημαντικά τα θέματα εκτέλεσης των μέτρων. Γιατί στη στρατηγική για την Βαλτική θάλασσα έχουμε μια εξαιρετική κατάσταση ουσιαστικά. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, οδηγίες, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά έχουν καταρτιστεί, έχουν ε, δημοσιευτεί, έχουν ε, γίνει υποδεκτά και τα κρατημέλη έχουν δεσμευτεί από νομικής άποψης. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να αξιοποιήσουμε την οδηγία για τα ύδατα ή για παράδειγμα να χρησιμοποιήσουμε την οδηγία για τις χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται δεσμευτικές ε, διατάξεις. Αναφέρεται όμως ότι και η γεωργία ως τώρα αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ε, Βαλτική θάλασσα. Προκαλεί προβλήματα στη Βαλτική θάλασσα, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει τα σχετικά και τα απαραίτητα μέτρα για να χρησιμοποιηθούν καλύτερα τα ήδη υφιστάμενα μέτρα. Θα πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση και της αλλιευτικής πολιτικής για να εγγυηθούμε την βιωσιμότητα της αλληλείας και σε ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις αλλιεύσης θα πρέπει να ανταποκρινόμαστε στις διεθνείς απαιτήσει. Άρα, αυτό που μας απασχολεί εμάς είναι η γεωργική γεωργία και η αλία για την διάσωση της Βαλτικής θάλασσας. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να αναφέρετε κάπου αυτό στην έκθεση. Σε ό,τι αφορά τα... Ε, φατουχάλατα. Ένα, μία από τις χώρες της Βαλτικής, η Σουηδία, έχει περάσει σχετική απαγόρευση. Θα ήταν σημαντικό να συμμετάσχουν και άλλα κράτη-μέλη. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό για το μέλλον της Βαλτικής και αυτό θα ήθελα να αναφέρετε στην έκθεση λοιπόν. Τώρα, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Nord Stream. Χαίρομαι που η συγκήτρια αποφάσισε να θέξει το θέμα αυτό. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίσουμε τις ενδεχόμενες συνέπειες ενός τέτοιου τεράστιου project στην περιοχή. Θα ήθελα ωστόσο να αναφέρεται ρητά στο κείμενο ότι το North Stream Ε, μπορεί να είναι, αν θέλετε, υπεύθυνο για να αποτραπούν περιβαλλοντικές συνέπειες. Αναφέρεστε βέβαια στο κείμενο σε αυτό, αλλά θα ήθελα να αναφέρεστε πιο ρητά. Για παράδειγμα, επειδή η εταιρεία θα αναλάβει τα έξοδα για την ε, διόρθωση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Και αυτό αποτελεί όρο που έχουν θέσει οι εμπλεκόμενες χώρες για την πραγματοποίηση του έργου αυτού. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναφερθεί αυτό από την εισηγήτρια. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι για το μέλλον της Βαλτικής ε, θα ήταν χρήσιμο να φροντίσουμε στο υψηλό επίπεδο, σε επίπεδο αρχηγός κυβερνήσεων, να συζητηθεί το θέμα. Γιατί αυτό, αν θέλετε, θα δώσει και πραγματική υπόσταση στα εφιστάμενα μέτρα. Σε ό,τι αφορά την αλία, τη γεωργία, την, ε, τον Stream, την ευθύνη των αρχηγών κυβερνήσεων. Όλα αυτά θα ήθελα να αναφερθούν, αν θέλετε, και τα χάλακτα. Ευχαριστούμε λοιπόν την εισηγήτρια. Ίσως να αναφερθούν και τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ που θα διατεθούν για τις ε, χώρες εκτός της Ένωσης. Συγγνώμη, τα 20 εκατομμύρια. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα, αυτά τα κονδύλια. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Μας θέσατε, στην... Ε, μας θέσατε και άλλα θέματα που είναι σημαντικά για την στρατηγική της Βαλτικής θάλασσας. Ο κύριος Πρόντι. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, μακροπεριοχές όπως τις κατονομάζουμε και αυτό είναι ύψης της σημασίας διότι και η κοινοπολιτεία ανεξαρτήτων κρατών μπορεί να αναμειχθεί, η Ρωσία δηλαδή. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πολιτική γειτονίας για τη συνεργασία με την ΚΑΚ. Γι' αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα των μακροπεριφερειών. Βεβαίως από ε, περιβαλλοντικής πλευράς η Βαλτική θάλασσα χαρακτηρίζεται από χαμηλό δίκτυ αλλαγών. Άρα από περιβαλλοντικής πλευράς πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο είναι εξαιρετικά ευάλωτο και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και αυτό αφορά ιδιαίτερα τα ποτάμια τα οποία εκβάλλουν στη Βαλτική θάλασσα. Νομίζω ότι η διευθέτηση αυτή θα πρέπει να επεκταθεί και σε όλες τις χώρες τις οποίες διατρέχουν αυτά τα ποτάμια. Είναι θέμα ύψης της σημασίας από περιβαλλοντικής πλευράς, δηλαδή οι μακροπεριφέρειες όπως τις κατονομάζουμε, θα πρέπει να είναι σε θέση να ορίζουν ε, ειδικέ σχέσεις, να προδιαγράφουν ειδικέ σχέσεις με άλλες μακροπεριφέρειες με τις οποίες γυτνιάζουν. Και αυτό έχει σχέση και με τον γεωργικό τομέα, ο οποίος επιδρά επί του υδροφόρου ορίζοντα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη Βαλτική. Πρόκειται για ζητήματα πολύ σημαντικά, τονίζω, αυτό το θέμα των μακροπεριφερειών, διότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά για ιδιάζοντα προβλήματα και νομίζω ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγι στην κατάσταση.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 Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια άλλη πτυχή του θέματος που συσχετίζεται με την ε, προστασία περιβάλλοντος. Θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα θέμα ε, ιστορικής σημασίας. Πρόκειται για τα χημικά όπλα τα οποία βρίσκονται στο βυθό της Βαλτικής μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα χημικά όπλα, τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα. Υπάρχουν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίσκονται στο βυθό της Βαλτικής και μπορεί να αποτελέσουν ένα ε, θέμα, μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ επικίνδυνο θέμα για το μέλλον αλλά και είναι Πότε θα μας απασχολήσει αυτό το θέμα, σε 10-20 χρόνια. Θα έπρεπε να προβλέψουμε συγκεκριμένες δράσεις για να δούμε τι εκπομπές προέρχονται από αυτά τα χημικά όπλα και τι επιπτώσεις υπάρχουν στον τομέα της αλίας. Ήδη αναφέρθηκαν προβλήματα στην Πολωνία, στον τομέα της αλίας εξαιτίας αυτών των χημικών όπλων το σημείο εκκίνησης θα πρέπει να αφορά την πρόσβαση στα στρατιωτικά αρχεία, να ξέρουμε για τι ποσότητες πρόκειται και να ξέρουμε πώς έχει η διάσταση αυτού του ζήτηματος. Είναι πολύ δύσκολο να αποτιμήσουμε το ζήτημα χωρίς να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Πράγματι, πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά ε, πάρα πολλέ λεκτηριόλες ουσίε εκεί και είναι ένα κίνδυνο ε, δεχόμενος, δεν έχει κανένα άλλος ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Άντερ Λίντον από την Εκτελεστική Επιτροπή έχει ζητήσει το, μπορεί να πάρει το λόγο και μετά στο τέλος η συγγήτρια. Ε, Ευχαριστώ για την επικοδομητική αυτή συζήτηση και τις πολλές πληροφορίες που ανέκυψαν από τη συζήτηση αυτή από τα μέλη της Επιτροπής. Από πλευράς Κομισιόν θεωρούμε ότι και η Επιτροπή Ρέτζι και η ΕΜΒΗ θα πρέπει να ασχοληθούν με αυτή την στρατηγική, την μακροοικονομική στρατηγική γιατί μας ενδιαφέρει το καλό input και η συνεχής πολιτική πίεση όπως είπε και ο Σουηδός συνάδελφος, θα πρέπει να είναι θέμα ύψης της προτεραιότητας και θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα σε πολιτικό επίπεδο αναμένουμε τη τελική έκδοση του κειμένου για να ενσωματωθεί στη στρατηγική μας. Η στρατηγική συνεχώς ενημερώνεται και επικαιροποιείται από ένα τέτοιο input και σας ευχαριστούμε για αυτή την εργασία. Ελπίζουμε να συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Ευχαριστώ, να Ράσπαχ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Αυτό που έχει σημασία είναι να συλλέξουμε όλες αυτές τις ε, προτάσεις για την αλλιευτική πολιτική, για τα φωσφορικά άλατα, για τα υπολείμματα, τα χημικά όπλα, όλα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα σφαιρικό πλαίσιο. Θα δω κατά πόσο μπορώ να ενσωματώσω αυτές τις προτάσεις τροπολογίες. Θα ήθελα όμως να έχουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσης και συμφωνώ με αυτά που είπαν όσοι παρενέβησαν. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς ε, μεταχειριζόμαστε τα υπολοιματικά ε, ύδατα, ε, τα απόβλητα από τα μεγάλα αστικά κέντρα, όλα αυτά τα οποία δεν πρέπει να εισραίουν στη Βαλτική θάλασσα. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να γίνει λόγος για το Δούναβι και άλλες θαλάσσιες ζώνες. Θα προσπαθήσουμε να τα ενσωματώσουμε όλα αυτά υπό μορφή τροπολογιών. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να αναβάλουμε την ε, υποβολή τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ για την εργασία σας. Πράγματι, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών λήγει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Πόσο γρήγορα πρέπει να δράσουμε για να μπορέσουμε έγκαιρα να ψηφίσουμε πριν από την Περιφερειακή Επιτροπή για να μπορέσει να ληφθεί υπόψη τη μας μελώνηση ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή μας στις 7 Απριλίου. Äh, Περνάμε στο σημείο 5 τη μερικής διάταξης. Προφορική ερώτηση του Chris Davis σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2053 για το οχήματα στο τέλος κύκλου ζωή του κατά τη χρονική περίοδο 2005-2008. Θα δώσω το λόγο στον Chris Davis για την ερώτηση και στην Κομισιόν μετά για να απαντήσει. Thank you, Chairman. Uh, Ευχαριστώ. Εν είδη εισαγωγή θα υποβάλω το ερώτημα στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης και θα ήθελα η Επιτροπή να απαντήσει πριν υποβάλω εγώ συμπληρωματική ερώτηση. Πράγματι μπορούμε όλοι να διαβάσουμε. Η Κομισιόν μπορεί να απαντήσει. Ο κύριος Κιούκλερ. Από την ίδια Ευσενλή ή όχι. Α, η κυρία Μπλάνκο. Παρακαλώ. Mr. Chair, good Καλό σας απόγευμα. Είμαι η κυρία Μπλάνκο από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Το ερώτημα του βουλευτή είναι κατά πόσο μπορεί η Επιτροπή να πει πώς ε, εφαρμόζεται η οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και κατά πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο αυτό. Θα ήθελα να τονίσω ότι πρόκειται για μία νέα προτεραιότητες Επιτροπής, δηλαδή να βελτιώσουμε την εφαρμογή, την τάχιστη εφαρμογή της οδηγίας. Πρόκειται για μια οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, όπου ε, θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένα νομικά μέσα για εφαρμογή αυτής της οδηγίας και αφήνουμε στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών ως προς τον τρόπο που θα εφαρμόσουν αυτή την οδηγία. Μία από τις βασικές προκλήσεις για την Επιτροπή, για την εφαρμογή της οδηγίας, αφορά το γεγονός ότι πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες ασχολούνται ως προς διαφορετικές πτυχές εφαρμογής, ε, περιφερειακές αρχές, ε, Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργεία Μεταφορών, Υπουργεία Περιβάλλοντος, όλα εμπλέκονται στην εφαρμογή της οδηγίας. Γι' αυτό η οδηγία, η εφαρμογή της ήταν δύσκολη και αν και έχουν επέλθει βελτιώσεις, η Επιτροπή πιστεύει ότι η οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής δεν έχει φτάσει στα οικονομικά και περιβαλλοντικά ωφέλη στα οποία θα έπρεπε να έχει φτάσει. Οι εξαγωγές οχημάτων τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, δηλαδή πολλούνται σε δεύτερο χέρι και που βρίσκονται στην ουσία στο τέλος του κύκλου ζωής, είναι ένα παράδειγμα της κακής εφαρμογής ε, και κακής ισχύω αυτής της οδηγίας, οδηγώντας σε απώλεια οικονομικών και περιβαλλοντικών ε, δυνατοτήτων. Πέρσι, τον Νοεμβρίου, η Επιτροπή ενέκρινε ένα έγγραφο για την εφαρμογή της οδηγίας για την περίοδο 2005-2008. Εδώ βλέπετε διάφορες δηλώσεις της Επιτροπής. σελίδα 1 μπορείτε να διαβάσετε ότι η έκθεση δεν ήταν ικανοποιητική. Στη σελίδα 2 η ποιότητα των, ε, των ποιοτικών προδιαγραφών είναι αμφισβητήσιμη. Η σελίδα 6, η συνολική ε, εφαρμογή θα πρέπει να βελτιωθεί. Αυτή είναι η τρέχουσα κατάσταση. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν σημαίνει ότι τώρα δεν έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Καταρχήν, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη σωστή μεταφορά της οδηγίας και υπ' αυτή την έννοια μπορώ να σας πω ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει ε, καθαρά νομικής φύσης ε, ε, μέτρα, δηλαδή έχει κάνει προσφυγή επί παραλήψη σε 14 περιπτώσεις, δύο υποθέσεις υπάρχουν ενώπιον του ΔΕΚ. Αυτή είναι η κατάσταση στο νομικό, ως προς το νομικό μέτωπο. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι κατευθυντήρες γραμμές έχουμε αναλάβει για να βελτιώσουμε την εφαρμογή της οδηγίας. Υπάρχουν δύο στόχοι για τα οχήματα στο τέλος ε, κύκλου ζωής, να μην ε, υπάρχουν πολλά ε, απόβλητα, δηλαδή να γίνεται ανακύκλωση εξαρτημάτων και ελπίζουμε τα κράτη-μέλη να φτάσουν στους στόχους, δηλαδή πρέπει να αποστέλουν πληροφορίες μέσω ερωτηματολογίου προς την Κομισιόν Υπάρχει δεσμευτική απογραφή που έγινε το 2008 για τα στοιχεία του 2006 και βλέπουμε σε αυτή την έκθεση ότι 13 κράτη-μέλη απέτυχαν στο, ως προς τους στόχους του 2006. Στη δεύτερη έκθεση που αφορά το 2007 βλέπουμε μία καλύτερη ε, απόδοση και το 2010, τώρα τον Ιούνιο, θα πρέπει να δούμε τα στοιχεία που αντιστοιχούν στο 2008. Ε, έχει επέλθει βελτίωση, αλλά όχι μέσα στα πλαίσια της αναμενόμενης πρόοδου. Ρωτήσαμε τα κράτη-μέλη να μας επεξηγήσουν την κατάσταση και τώρα ε, αναλύουμε τις απαντήσεις που λάβαμε. Θα ήθελα να σας πω ότι στις απαντήσεις που εξετάσαμε, οι λόγοι που προβάλλουν τα κράτη-μέλη αφορούν καθυστερήσεις έτσι ώστε να είναι υπόλογοι οι οικονομικοί εμπλεκόμενοι φορείς σε σχέση με τα εξαρτήματα. Οι οικονομικοί φορείς από ασφαλιστικές εταιρείες, εισαγωγής, εξαγωγής, και ούτω καθεξής ασχολούνται, όλοι αυτοί εμπλέκονται ε, σε αυτή την οδηγία. Τα κράτη-μέλη επίσης προβάλλουν το γεγονό ότι δεν υπάρχουν μέσα παροπλισμού. Ίσως θα πρέπει να συντάξουμε και τις δύο πλευρές των απαντήσεων, αυτά σε σχέση με την εφαρμογή. Μετά τις διαφορές που είδαμε κατά την αποτίμηση των εθνικών εκθέσεων, φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι δεν αποτελούν το τέλος της ιστορίας και ίσως η αποτυχία της συνολικής εφαρμογής της οδηγίας ε, ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογίες για να ανταποκριθούν στους στόχους της οδηγίας. Άρα για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δυσκολία και για να φτάσουμε σε μια κοινή μεθοδολογία για την αποτίμηση των στοχοθετήσεων, έχουμε προβεί στη σύσταση μιας ομάδας εργασίας σε σχέση με τη μεθοδολογία, έτσι ώστε να συντάξουμε κοινές κατευθυντήριες γραμμές. Αυτή η ομάδα εργασίας απαρτίζεται όχι μόνο από τα κράτη-μέλη, αλλά και από εκπροσώπους του βιομηχανικού κλάδου. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία διότι ο βιομηχανικός ε, κλάδος είναι υπεύθυνο για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Ένα άλλο σημείο που σχετίζεται με την κακή εφαρμογή σχετίζεται με το σύστημα διαχείρισης γενικότερα που ισχύει στα κράτη-μέλη. Πέρσι το Δεκέμβριο η Επιτροπή απέστειλε ένα ερωτηματολόγιο σε όλα τα κράτη-μέλη ζητώντας τα συνολικά στοιχεία αποτίμησης των οχημάτων αυτών. Δηλαδή πόσο οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι, τον αριθμό οχημάτων, εισαγωγές, εξαγωγές και ούτω καθεξής και ε, στην Επιτροπή ε, Τεχνικών Προσαρμογών συζητάμε το θέμα εξαγωγών ε, ήδη χρησιμοποιημένων οχημάτων. Ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να υποβάλουν στην Επιτροπή αριθμητικά στοιχεία για τα εξαγόμενα οχήματα και τις χώρες προορισμού και αναμένουμε αυτά τα στοιχεία έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να προβούμε σε περαιτέρω ανάλυση. Τι άλλο μπορεί να γίνει στο μέλλον. Γιατί μέχρι τώρα σας είπα ποια είναι τα μέτρα που έχουμε αναλάβει. Ένα μέτρο που συζητείται με τα κράτη-μέλη είναι το κατά πόσο πρέπει να τροποποιήσουμε το ερωτηματολόγιο της οδηγίας για τις τριετής εκθέσεις. Αυτό το λαμβάνουμε υπόψη, το εξετάζουμε. Ένα άλλο ε, ενδεχόμενο ζήτημα που συζητάμε στην ομάδα εργασίας με τα κράτη-μέλη είναι κατά πόσο θα ε, πρέπει να εισαγάγουμε τροποποίηση στον τρόπο ε, ετήσιας παροχής στοιχείων. Εάν οι κατευθυντηρίες γραμμές δεν επαρκούν και τέλος θα ήθελα να σας πω ότι η Επιτροπή για όλα τα θέματα περιβάλλοντος που σχετίζονται με τον τομέα ε, τονίζω ότι θα πρέπει να γίνονται επιθεωρήσεις της οδηγίας για τα απόβλητα. Έχουμε προβεί σε μία μελέτη αντικτύπου για θετική αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον εάν προβάλλουμε αυτά τα μέτρα. Άρα συνεχίζουμε με αυτή την ε, προοπτική και για να συνοψίσω, κύριε Ντέιβις, αγαπητά μέλη, η Επιτροπή δεν είναι ικανοποιημένη από την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία βρίσκονται εν εξελίξη στη συνεργασία με το τομέα αυτοκινητοβιομηχανίας. Θα θέλαμε όμως να συνεργαστούμε μαζί σας έτσι ώστε οι αλλαγές να επέλθουν πολύ νωρίτερα από ό,τι είδαμε τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο Κρίς Ντέιβις. Ευχαριστώ. Εδώ και 10 χρόνια η οδηγία έχει τεθεί ισχύ, γι' αυτό θα πρέπει να αποτιμήσουμε την κατάσταση. Μιλάμε για 25 με 30 εκατομμύρια οχήματα τα οποία έχουν παροπληστεί Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ε, νομοθεσία έτσι ώστε ο Μολύνων να καταβάλει το αντίτιμο και να, γίνονται, να γίνεται και ανακύκλωση ε, στην περίπτωση, στις περιπτώσεις αυτές των οχημάτων που παραπλήσονται. Γιατί πολλά οχήματα μπορούν να ανακυκλωθούν στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την αποτίμηση της κατάστασης. Στις συζητήσεις που είχαμε με την Επιτροπή και στο Ηνωμένο Βασίλειο βλέπω ότι η Επιτροπή ασχολείται με τις στοχοθετήσεις, κατά πόσο δηλαδή έχουμε ανταποκριθεί. Σε μερικά κράτη-μέλη υπάρχουν καλά αποτελέσματα. Χρειαζόσαστε όμως ακριβείς πληροφορίες για τον συνολικό αριθμό οχημάτων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Αν δούμε τα στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου, Πιστεύω ότι παίρνετε ένα 50% των συνολικών στοιχείων που χρειάζεστε. Άρα η ανάλυση σας είναι μεροληπτική. Είναι ελληματική γιατί δεν έχετε όλα τα στοιχεία. Υπάρχει έλλειψη πολιτικής θέλησης για να εφαρμοστεί η νομοθεσία σε ορισμένα κράτη-μέλη και σε ορισμένα κράτη-μέλη καταδεικνύεται πολύ καλά ε, η κατάσταση Σουηδία, Ολλανδία, Δανία. Η κατάσταση εκεί είναι εντελώς διαφορετική. Γι' αυτό αναρωτιέμαι γιατί η Επίτροπη δεν ε, επιβάλλει στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος τέτοια θέματα στην ατζέντα δηλαδή των Υπουργών έτσι ώστε να μας πείτε ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι οι κακοί μαθητές έτσι ώστε η κάθε κυβέρνηση να γυρίσει πίσω και να πει στους δημοσίους υπαλλήλου προσέξτε περισσότερο γιατί δεν θέλω να έρθω σε αυτή τη δύσκολη θέση ξανά. Γιατί σε κανέναν δεν αρέσει αυτό και ίσως θα έπρεπε να φυγεί κατά αυτόν τον τρόπο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ένα ιδιάζον θέμα που ίσως αφορά και άλλα κράτη. Έχουμε την Επιτροπή ε, μητρών Καταγραφής Οχημάτων με βάση τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου υπάρχουν σαφή μητρώα. Δεν έχει κίνητρα ή δεν, δεν έχουν δοθεί οδηγίες σωστές για να ανταποκριθεί ως προς αυτά τα οχήματα είναι η πιο ε, γραφειοκρατική οργάνωση που έχω γνωρίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία από τις πιο γραφειοκρατικές. Αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην νομοθεσία, όταν όχημα φτάσει στο, τέλος κύκλου ζωής, τότε θα πρέπει να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό διάλυσης. Όμως υπάρχει ένα παραθυράκι εδώ. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ θα το κάνω αυτό. Δηλαδή βάζεται ένα χ σε ένα τετραγωνίδιο που λέει ότι ο υποφαινόμενος θα καταστρέψει το όχημα και άρα δεν απομακρύνεται από τα μητρώα. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν φεύγει από τα μητρώα, αλλά στην ουσία διαλύεται, υποτίθεται. Πολλά από αυτά τα οχήματα πάνε στην ε, πρώην Ανατολική Ευρώπη. Ποιος είναι υπόλογος για αυτά. Πολλά από αυτά ίσως ξαναβρίσκονται στους δρόμους, τα οδηγούν εγκληματίες υποτίθεται ότι διαλύονται αλλά δεν βγαίνουν από τα Μητρώα. Άρα η Επιτροπή δεν μπορεί να έχει ακριβή στοιχεία. Αν λοιπόν η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει προσφυγή επί κατά της χώρας μου, τότε ε, θα σας πούν από το Ενωμένο Βασίλειο ότι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να ορίζει την απομάκρυνση από τα Μητρώα την, ε, δηλαδή, την διαγραφή από τα Μητρώα. Άρα θα σας πω από το Ηνωμένο Βασίλειο εμείς ακολουθούμε το γράμμα του νόμου. Αναρωτιέμαι λοιπόν κατά πόσο ε, θα πρέπει να αναδιατυπώσετε την ομοθεσία είτε να ορίσετε κατευθυντήριες γραμμές έτσι ώστε να κλείσουν αυτά τα παραθυράκια ή κάτι άλλο που θα μας πείτε εσείς. Ο Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ. Και θα να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Ντέιβις και την Επίτροπη. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος για να γίνει αναδιατύπωση ανάλογη με αυτή που αφορά τα απόβλητα των ε, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών. Θα έπρεπε να γίνει κάτι ανάλογο, διότι μιλάμε για ανάκτηση πόρων. Περισσότερο για ανάκτηση πόρων παρά για θέμα περιβάλλοντος. Θα πρέπει να γίνει μια επαναδιατύπωση της οδηγίας, ίσως έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ανάθεση ευθυνών και στο βιομηχανικό τομέα, την αυτοκινητοβιομηχανία διότι υπάρχει υπερπαραγωγή οχημάτων, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, και νομίζω ότι εν μέρη αυτές οι μονάδες θα έπρεπε να αφοσιωθούν στην καλύτερη διάλυση οχημάτων, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει πιο επιλεκτική ανακύκλωση είτε εξαρτημάτων αλλά και υλικού γενικότερα. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν οι δύο αντίποδες και μέσα σε αυτούς δύο πόλους, εν πρέπει να γίνει αναδιατύπωση. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστώ την ε, Κομισιόν για τις ανοιχτές ερωτήσεις που μας, απαντήσεις που μας έδωσε. Νομίζω ότι αναφέρθηκε πραγματικά στα πρακτικά προβλήματα που υπάρχουν κατά την εφαρμογή αυτή τη οδηγία, η οποία ξεκίνησε με καλές προθέσει, αλλά οδήγησε σε πολλά προβλήματα όταν πρόκειται να εφαρμοστεί σωστά. Αυτή είναι τώρα η μεγάλη πρόκληση για μας. Να βρούμε δηλαδή τις ε, δυνατότητες για να την ε, καταστήσουμε λειτουργική στην πράξη. Υπάρχει καλή πρόθεση. Αλλά πολλοί αναρωτιόνται πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη. Και θα πρέπει η Κομισιόν ε, να φροντίσει να ξανασκεφτεί αυτές τις πτυχές, γιατί από την απάντηση της Κομισιόν είδαμε ξεκάθαρα ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα εφαρμογής και ότι δεν υπάρχουν καν κατευθυντήριες γραμμές, πράγμα που με κάνει να απορώ πάρα πολύ, γιατί η οδηγία αυτή χρονολογείται από το 2000 και το σύστημα δεν πολύ λειτουργεί. Γι' αυτό θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας να δούμε τι θα κάνουμε για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που έχουμε όσον αφορά την έννοια του Ευρωπαίου κατασκευαστή κλπ. κλπ. Γιατί είναι δικαιολογημένες νομίζω οι παρατηρήσεις που γίνονται και θα ήθελα να παρακαλέσω την πρόσωπο της Κομισιόν να μας πει ποιε είναι οι σκέψεις που υπάρχουν στην Κομισιόν τώρα ούτω ώστε αφενός αυτό το υλικό που χρειάζεται ακόμα, Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και που υπάρχει στα παλιά αυτοκίνητα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από την άλλη μεριά τα αυτοκίνητα να μην πετιώνται κάπου αλλά να προωθούν σε μια οργανωμένη διάλυση ή να για να χρησιμοποιηθεί το υλικό που περιέχουν, πράγμα που έχει και οικολογική σημασία. Δεν μπορούμε να λέμε τα κράτη-μέλη δεν δίνουν αρκετά στοιχεία. Περιμένει η Κομισιό να κάνει προτάσεις τι θα πρέπει να γίνει ούτω ώστε να μπορούμε να βασιζόμαστε καλύτερα στα στοιχεία αυτά. Δεν μπορούμε να φιόμαστε στα κράτη-μέλη. Δεν είναι σωστό αυτό γιατί αν τα κράτη-μέλη δεν θέλουν δεν θα κάνουν κάτι παραπάνω από εκείνο που είναι απόλυτα υποχρεωμένοι να κάνουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντέιβις. Γιατί το πρόβλημα που συζητάμε αυτή τη στιγμή δεν είναι καινούριο πρόβλημα, δεν είναι ένα θέμα που μόλις αρχίζουμε να συζητάμε. Από ό,τι κατάλαβα χρειαζόμαστε πληροφορίες για την εφαρμογή της οδηγίας ε, στο παρελθόν, δηλαδή μεταξύ του 2005 και 2008. Και σήμερα βρισκόμαστε στο 2010. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον αυτή η οδηγία εφαρμόζεται και πώς εφαρμόζεται. Από ό,τι ακούσαμε και από την Κομισιόν υπάρχουν προβλήματα κατά την εφαρμογή της οδηγίας σε κράτη-μέλη. Η κυρία Διευθύντρια ανέφερα ότι το ίμιση περίπου των κρατών μελών δεν έχουν καθόλου εφαρμόσει σωστά αυτή την νομοθετική πράξη. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποια πειθαρχία θα έλεγα. Αυτές οι χώρες που δεν έχουν εφαρμόσει την οδηγία θα πρέπει να τύχουν κυρώσεων. Και αυτό που είναι λυπηρό επίσης είναι να ακούμε ότι καθυστερείται η εφαρμογή της οδηγίας λόγω της έλλειψης βούλησης των ελόγων κρατών μελών. Εγώ δεν ε, μπορώ να φανταστώ ότι κάποιοι όμως δεν μπορούν, θέλουν να εμπλακούν εδώ στον οικονομικό τομέα. Ίσως ορισμένες άλλες οδηγίες παρεμποδίζουν τη σωστή λειτουργία αυτών των οικονομικών παραγόντων. Θα πρέπει να το εξάσουμε και από αυτή τη σκοπιά για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτές τις μονάδες όπου μπορούν να προσφέρονται αυτές οι υπηρεσίες για τα οχήματα που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπως και ο κύριος Ντεβίς θα ήθελα και εγώ να έχω πληροφορίες πού βρίσκονται ακριβώς τα προβλήματα και πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε. γιατί μπορούμε βέβαια να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη με κάποια πίεση να φροντίσουν η οδηγία αυτή να εφαρμόζεται σωστά. Όταν εγώ ήμουν στην Πολωνία, ε, στην Εθνική Βουλή, συνεργάστηκα για την εφαρμογή της οδηγίας και ήμασταν σίγουροι ότι τα πράγματα θα πήγαιναν σωστά. Αλλά όταν μας λέει τώρα η Κομισιόν ότι υπάρχουν κράτη-μέλη στα οποία δεν εφαρμόζει σωστά η οδηγία αυτή, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι αυτά τα κράτη-μέλη. Για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν θέλει κανένα άλλο το λόγο, οπότε θα μπορούσα να δώσω το λόγο πάλι στην Κομισιόν. Παρακαλώ, η φαίνεται κύριε Μπλάνκο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Άκουσα προσεκτικά αυτά που είπαν οι εξώτιμοι κύριοι κύριοι βουλευτές και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω που είπαν ότι η έκθεσή μου ήταν τίμια βέβαια, ήταν πάρα πολύ τίμια, σωστή και έχω να σα πω ότι η Κομισιόν εργάστηκε σκληρά με τα κράτη-μέλη και με την βιομηχανία για να μπορέσει να εφαρμοστεί η οδηγία αυτή σωστά. Είναι αληθέα ότι η κατάσταση δεν είναι ακόμα πλήρω ικανοποιητική. Θα ήθελα όμω να τονίσω ότι βελτιώνεται σιγά-σιγά. Επιλέξαμε αυτή την ε, μέθοδο βελτίωσης των αποτελεσμάτων με συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και όπως είπα αρχικά αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε ένα σημαντικό έγγραφο που μπορεί να εγκριθεί από, την, ε, από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο μέσα στα πλαίσια της ένα που μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο κατά το γνώμη μου παραδείγματος χάρη ένας θέμα της εξαγωγής ε, των αποβλήτων των οχημάτων ή της εξαγωγής των παλαιών οχημάτων. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούμε να τα θεωρήσουμε σαν απορρίμματα και να ελέγχονται κατά τον ίδιο τρόπο όποιο οποιαδήποτε άλλη μεταφορά αυτού του τύπου. Από ό,τι ακούσαμε με διάφορες φαίνεται ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε πιο ριζοσπαστική αντιμετώπιση και να τροποποιήσουμε την οδηγία. Όμως, έχει αφαιθεί στην διακριτική ευθεία των κρατών μελών να αποφασίσουν πώς θα ε, μεταφέρουν και θα εφαρμόσουν την οδηγία αυτή σε ορισμένε χώρε χρειάζεται αυτό το πιστοποιητικό διάλυση που να το υποβάλλεται στι αρχέ εάν θέλουν να σταματήσουν να πληρώνουν τον φόρο τα δέλη μάλλον κυκλοφορία. Εκεί λειτουργεί πράγματι το σύστημα. Γιατί αν δεν έχει κανένα αυτό το πιστοποιητικό διάλυση του οχήματο που το εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές εξακολουθεί κανένα να είναι υποχρεωμένο να καταβάλει τα τέλη κυκλοφορία. Αυτό δεν σημαίνει όμως παντού. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει και το Ιούνιο θα δούμε αμέσως ε, κατά πόσον έχει βελτιωθεί η απόδοση της εφαρμογής. Εάν όχι, θα πρέπει να αξιολογήσουμε και άλλες δυνατότητες που ίσως συμπεριλαμβάνουν και τη δυνατότητα να ξαναδιατυπωθεί η οδηγία, να καταστεί πιο αυστηρή, να υπάρχουν άλλες διατάξεις κλπ. Και θα πρέπει να επανέλθω εδώ μετά που θα έχω τα αποτελέσματα αυτής της ε, επανεξέτασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Ντέιβις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν την απάντησή της. Είπε η εκπρόσωπος της Κομισιόν θα ξαναεξετάσει τα στοιχεία τον Ιούνιο. Και αν δεν υπάρχει σημαντική πρόοδος, μπορεί να ε, υιοθετήσει κάποιες από τις ριζοσπαστικές ε, προτάσεις που προτείναμε. Δεν ξεχνάμε, η Κομισιόν έχει το δικαίωμα πρωτοβουλία, αλλά οι βουλευτέ συμφωνούν μαζί μου να επανέλθουμε αργότερα για να δούμε ποια είναι η αξιολόγηση που έχει κάνει η Κομισιόν τη όλη κατάσταση. Το σημειώνουμε, λέει ο Πρόεδρος. Και περνάμε στο άλλο σημείο σήμερα τη διάταξη. Προφορική ερώτηση για τα κριτήρια εφορία των βιοκαυσίμων. Έχει υποβληθεί από του κυρίου Έκχαουτ, Αρσένη Λάνζ και και Λεπάζ. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Έκχαουτ, εάν θέλει κάτι να σχολιάσει, να δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν. Ναι, δύο λόγια, Πρόεδρε. Η ερώτηση είναι πολύ σαφής νομίζω. Θα ήθελα βέβαια να τονίσω ότι από τότε που υποβάλαμε την ερώτηση αυτή άλλαξαν κάποια πράγματα στην τρίτη ερώτηση παραδείγματο χάρη που ρωτάμε ποια είναι η θέση όσον αφορά τα κριτήρια εφορία για τα βιοκάστημα και τη βιομάζα. Ξέρουμε τώρα την απάντηση, δεν χρειάζεται να επισέλθω τι λεπτομέρειε. Και επίσης δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε εδώ δεσμευτικά κριτήρια. Το θέμα των κριτηρίων αηφορίας για το βιοκαύσιμα και τη βιομάζα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είχαμε έντονη συζήτηση την περασμένη θητεία με την Κομισιόν. Ε, τώρα έχουμε νέο κοινοβούλιο, νέα εκτελεστική επιτροπή, νέους επιτρόπους τουλάχιστον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δώστε μας μια σύνομη απάντηση στα τρία θέματα. Πρώτον, όσον αφορά την εφαρμογή των κριτήριων αειφορίας. ιδίω τον ορισμό των συνεχώς δασωμένων περιοχών που είναι περίεργη γιατί μπορεί να οδηγήσει παραδείγματο χάνει σε αποψήλωση φυτίων φοινικοδέντρων κλπ. Είναι δύσκολο. Το δεύτερο, όσον αφορά την έμεση χρήση των γιών, γιατί ξέρει η Κομισιόν υπάρχει το πρόβλημα της έμεις αλλαγής χρήσης της γης για τη βιομάζα και τέλος το τελευταίο σημείο όσον αφορά τα κριτήρια εφορίας για την βιομάζα όσον αφορά τα κράτη-μέλη και την σχετική βιομηχανία. Πρώτα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Έχουμε και από τις δύο γενικές διευθύνσεις εκπροσώπους, ενέργεια και κλίμα. Ο κύριος Μπαμπάσο από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας θα πάρει το λόγο. Κύριος Μπαμπάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στις τρεις ερωτήσεις που το βλήθησαν. Η μία που αφορά τα κριτήρια εφορίας για τα βιοκαύσιμα και τη βιομάζα γενικά. Οι κύριοι βουλευτές που να τις ερωτήσεις αυτές συγκέντρωσαν την προσοχή τους σε ένα από τα κριτήρια αηφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα υγρά βιοκαύσιμα. Εμείς από πλευράς Κομισιόν θα ήθελα να σας πω ότι το σχέδιο αηφορίας θα πρέπει να εξασθεί σε ένα σύνολο βιοκαύσιμα και βιομάζα θα πρέπει να ακολουθούν όλα τα κριτήρια για να μπορούν να συμπεριληφθούν. Τα διάφορα κριτήρια που αφορούν την εξοικονόμηση των ε, αερίων του θερμοκηπίου και ε, γη τις οποίες η χρήση αλλάζει και γη η οποία αποθηκεύει μεγάλες ε, ποσότητες άνθρακα, όλα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν από κοινό. Εξετάζουν λοιπόν όλα τα κριτήρια μαζί, η Κομισιόν δεν βλέπει πώς η μετατροπή των τροπικών δασών σε φυτίες φοινικοδέντρων θα μπορούσαν να είναι συμβατές με τα κριτήρια. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτηση που αφορά τις έμεσες αλλαγές της χρήσης της γης, Αρχίσαμε να εργαζόμαστε στο θέμα αυτό αμέσως μετά την υιοθέτηση της οδηγίας για τις ανώσιμες πηγές ενεργείας. Και εμείς τώρα, αυτή τη στιγμή, ε, βασιζόμαστε στις εξής αναλυτικές ε, μεθόδους. Η μία που βασίζεται σε ένα πρότυπο ισορροπίας που βασίζεται σε που εξετάζεται με υπολογιστές και το δεύτερο σε μερική ισορροπία του μοντέλου. Επίσης επανεξετάζουμε τη βιβλιογραφία. Παρ' όλα αυτά, έχω να σας πω ότι και στις πιο προχωρημένες από αυτές τις ε, δοκιμασίες αναγνωρίζεται ότι χρειάζεται και συμπληρωματική εργασία για να μπορούν να υποβληθούν ακριβείς συστάσεις για τους νομοθέτες η νομοθεσία προτι... προβλέπει η Κομισιόν εξτάσει το θέμα με υποβολή πρόταση ενδεχομένω μέχρι το Δεκέμβριο του 2010. Ελπίζω ότι μέχρι τότε θα έχουμε ολοκληρώσει την εργασία μας. Όσον αφορά το τελευταίο ερώτημα για την αηφορία της βιομάζας και τα σχετικά κριτήρια, ο εξώσιμος βουλευτή που πήρε το, λόγο τόνισε ότι μεταξύ η Εκτελεστική Επιτροπή υπέβαλε μια ανακοίνωση. Χρειαστήκαμε λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι είχε προβλεφθεί αρχικά, γιατί αποφάσισε η Κομισιόν να περιμένουμε να είναι λειτουργική η νέα Επιτροπή υπό τη νέα της δηλαδή σύνθεση και να μην αφήσουμε την εξερχόμενη Επιτροπή να υιοθετήσει την ανακοίνωση αυτή. Και μόλις όταν ανέλαβε τις υποχρεώσεις της στις 25 Φεβρουαρίου, η νέα επιτροπή στις 25 Φεβρουαρίου η Κομισιόν προετοίμασε μια δήλωση. Αυτή η έκθεση δεν προβλέπει ένα νομοθετικά θεσμευτικό σχέδιο αηφορίας, προτείνει όμως τα κριτήρια εφορία να χρησιμοποιηθούν από εκείνα τα κράτη-μέλη που θέλουν σε εθνικό επίπεδο να υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόγραμμα. Η Κομισιόν έλαβε υπόψη γνωμοδοτήσεις των εμπειρογνωμόνων αυτά που αναφέρουν στη βιβλιογραφία και μια έκθεση που έγινε επί τόπου και που στηρίζεται σε τρεις εξωτερικές εκθέσεις. Θα σας δώσω κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά αυτές τις δημόσιες διαβουλεύσεις, για τις οποίες πήραμε 252 απαντήσεις. Οι ερωτήσεις αφορούσαν πέντε κυρία θέματα. Το κατά πόσο χρειάζεται ένα σχέδιο εφορίας για τη βιομάζα. Δεύτερον, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ε, τρίτον, η πρόθεση της ε, αποδεσματικότητας της έμεσης αλλαγής χρήσης γης. Και τέλος είχαμε τα θέματα αξιολόγησης και ε, στην ιστοθελίδα ε, της Κομισιόν μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα αυτών των μελετών. Κατόπιν όλες αυτές τις προβαρισκευτικές εργασίες, η Κομισιόν εξέτασε όλες τις διαθέσιμες ε, δυνατότητες που υπήρχαν και είδε ποια είναι η ισορροπία με το ξύντο να υπάρχει συμπληρωματική επιβάλληση σε χιλιάδες παραγωγούς βιομάζας και βιοκαυσίμων και τις συμπληρωματικές ασφαλίσεις που θα μπορούσαν να υπάρχουν από ένα εναρμονισμένο σύστημα κριτηρίων αηφορίας για τη χρήση της βιομάζας. Ε, πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη θέλουν να υπάρχουν κριτήρια αηφορίας ε, για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα και τα περισσότερα κρατημέλη θεωρούν ότι υπάρχει ε, σωστή ισορροπία. Όχι μόνο γιατί η βιομάζα είναι ένας από τους κύριους φορείς για να πετύχουμε τους στόχους μας για την ανανεώσιμη ενέργεια. Αλλά εκτός αυτού εξετάζουμε όλα τα πράγματα αυτά συνεχώς και αυτό σημαίνει ότι σε ένα χρόνο θα ξανααξιολογήσουμε τα αποτελέσματα των συστάσεων και αν χρειαστεί θα ακολουθήσουμε διαφορετική άγουσα. Ευχαριστώ πολύ. Σα ε, Σας ευχαριστώ και έχουμε μαζί μας και ένα εκπρόσωπο από την ε, Γενική Διεύθυνση για το Κλίμα. Ο κύριος Owen, αν έχετε να προσθέσετε κάτι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος για να απαντήσω στα ερωτήματα. Να πω απλά ότι υπάρχει στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και τη δική μας διεύθυνση για τις ε, δράσεις για το περιβάλλον. Συζητάμε και υπάρχει έντονο διάλογος και υποστορίζω όλα όσα είπε ο προλαλή σα. Μου άρεσε αυτό που είπατε ότι σε κάποιες περιπτώσεις ο διάλογος είναι πιο έντονος από τις άλλες περιπτώσεις. Ο κύριος Πρόντι. E Ευχαριστώ τους συναδέλφους για το ερώτημα που υπέβαλαν στην Επιτροπή και νομίζω ότι εδώ γενικότερα θα πρέπει να συζητήσουμε τη συμβατότητα και τα ανταγωνιστικά πρότυπα των αρωτριέων γεών. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει μόνο η παραγωγή βιομάζας, αλλά καταβάλλεται πίεση για αλλαγή χρήσης γεών στην ε, γεωργία έτσι ώστε να παραχθεί φωτοβολταϊκή ενέργεια. Αυτό θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Δηλαδή γίνεται μία συζήτηση. Θα πρέπει μάλλον να γίνει το ταχύτερο δυνατόν για το θέμα των αρωτρίων γεών για σκοπούς παραγωγής τροφίμων ή ε, παραγωγής ενέργειας. Αυτό είναι θέμα πολύ λεπτό για πολλές χώρες, γιατί συμφωνούμε ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι η παραγωγή τροφίμων. Θα πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν το όλο ζήτημα. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να αρχίσουμε με την χρήση όλων των υπολοιμάτων, είτε γεωργικών είτε δασοκομικών, για να ορίσουμε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Και Στη συνέχεια υπάρχει ένα περιθώριο για να δοκιμάσουμε ε, ε, ενεργειακές καλλιέργειες σε μολυσμένες ε, γέες. Στην Ιταλία έχουμε ένα 3% μολυσμένων γεών και ίσως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Μιλάμε για 10.000 τετραγωνικά μέτρα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αρχίσουμε με αυτές τις ε, μολυσμένες γέες για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προβάλλουμε ε, καλλιέργειες ε, του ενεργειακού τομέα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε πόσος χρόνος θα χρειαστεί και γι' αυτό. Για να δούμε και το θέμα της συμβατότητας και της αλλαγής χρήσης γης ως προς τις ε, αρρώσιμες γης, δηλαδή κατά πόσο μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για παραγωγή τροφίμων ή για ενεργειακούς σκοπούς, όχι βιομάζα. θα σας ε, αναφέρω μια επιστολή 25 μη κυβερνητικών οργανώσεων που έστειλαν την προηγούμενη εβδομάδα στους αρμόδιους και στον πρόεδρο της Επιτροπής εκφράζοντας τις ανησυχίες τους σχετικά με την ε, πρακτική εφαρμογή των ευρωπαϊκών ε, κριτηρίων βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα και την βιομάζα. Συγκεκριμένα παρόλο που θύχτηκε το θέμα πριν ε, στην απάντηση, θα ήθελα να ζητήσω και πάλι ένα σχόλιο, μια και ζητούν ε, η Επιτροπή να αποκλείσει ότι οι, φε, οι φυτίες φοινικόδεντρων θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως συνεχώς δασωμένες περιοχές. Και ακόμη να διευκρινίσει ποια βιοκαύσιμα και τα υπολείμματα ή τα παράγωγά τους συμβάλλουν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, Mr. Σας ευχαριστώ. Thank you, Chairman. Um, I, I thank the Commission. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις απαντήσεις που μας έδωσε. Να πω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιεί πολλά λόγια και τελικά δεν μας λέει πολλά καινούργια στοιχεία, δεν μας παρουσιάζει πολλά καινούργια στοιχεία. Εγώ έχω μία ερώτηση να κάνω. Είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα υπάρξουν φυτίες φαινικόδαντρων σε ό,τι αφορά τα κριτήρια αηφορία σε περιπτώσεις που παλαιότερα υπήρχαν δάση. Τι σημαίνει αυτό το normal, υποκρανικές συνθήκες. Αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρξουν τέτοιες φυτίες φαινικόδοντρων που θα πληρούν τα κριτήρια αηφορίας ή εξακολουθούν να υπάρχουν παραθυράκια, αν θέλετε, τα οποία ενδεχομένως να περάσουν. Ευχαριστώ, κυρία Μακεβένα. Ναι, να πω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει ε, έντονο ενδιαφέρον από το κοινό για το θέμα αυτό και παρακολούθησα διάφορες συνεντεύξεις τύπου για την έκθεση αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι δύσκολο γιατί δεν την έχουμε δείξει στη τελική ανάλυση την ε, έκθεση αυτή την, της Επιτροπής. Πολλοί από τους εμπειριογνώμονες, αν θέλετε, ε, διατελούν σε καθεστώς σύγχυσης. Δεν βλέπουν να υπάρχει μια σαφή πρόταση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία από τις προτάσεις που έχω εγώ εδώ αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η μετατροπή δασωμένων περιοχών σε φυτίες φινικόπιτρων δεν αποτελεί απαραίτητα παραβίαση των κριτηρίων. Άρα έχω να σας πω την αλήθεια, μπερδευτεί. Τι θα γίνει δηλαδή, θα συνεχίσουν να υφίστανται οι υφιστάμενες οι φοιτίες, φαινικόδοντρων, αλλά θα δημιουργηθούν καινούριε. Αν θα θέλατε παρακαλώ να μου το διευκρινίσετε το θέμα αυτό, γιατί ξέρετε ενδιαφέρει ιδιαίτερα την επικράτειά μου και τον τύπο. Πότε θα δημοσιευθεί αυτή η έκθεση επίσης και τι θα ακολουθήσει μετά τη δημοσίευση της έκθεσης. Ο κύριος Eichhout, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πρώτες αυτές απαντήσεις, αλλά θα ήθελα να συμφωνήσω και εγώ με τους συναδέλφους ότι ως τώρα οι απαντήσεις αυτές δεν είναι τόσο σαφείς. Καταρχάς, για τα τρία θέματα. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τον ορισμό των φυτιών φοινικόδοντρων. Γιατί δεν ακολουθήσατε την, ε, τον ορισμό του ΦΑΟ, όπου γίνεται σαφής εξαίρεση για συστήματα αγροτικής παραγωγής, τα οποία δεν θεωρούνται ότι υπάγονται στην δασοκομεία. Ξέρω ότι υπάρχουν πιο πολλά κριτήρια, πιο πολλοί όροι στο έγγραφο, αλλά αν τώρα μιλάμε για δάση χαμηλής βιοπικιλότητας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, μπορεί να συμβεί εκεί τέτοια αλλαγή από δάσο σε φυτία και να θεωρηθεί ότι παρόλα αυτά είναι ε, αηφόρο το σύστημα αυτό. Εμείς θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να μην θεωρείται αηφόρος μια τέτοια μεταστροφή. Γιατί δεν ακολουθούμε λοιπόν την, ε, τον ορισμό του ΦΑΟ που είναι πολύ πιο σαφής. Τώρα, για την έμεση αλλαγή ε, γεών. Ξέρω τα μοντέλα που υπάρχουν. Γνωρίζω ποια είναι αυτά αλλά πολύ φοβάμαι ότι οι επιστήμονες ε, δεν ε, συμφωνούν ότι είναι σαφή τα μοντέλα αυτά, γιατί τα μοντέλα αυτά, αν θέλετε, θα πάντα αποτελούν μια απλοποίηση και μέχρι το τέλος του 2010 δεν θα καλύπτουν απόλυτα την πραγματική κατάσταση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι κανένα από αυτά τα μοντέλα δεν δείχνει ότι δεν υπάρχει καθόλου έμεση αλλαγή της χρήσης της γης. Άρα εκεί έρχεται και εφαρμόζονται και η αρχή της πρόληψης. Άρα, τι θα γίνει για να ληφθεί υπόψη το γεγονός αυτό. Μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώς τα ποσοστά, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Και κατά τρίτον, λέτε ότι η τρέχουσα ανακοίνωση για την βιομάζα έχει βρει τη σωστή ισορροπία και θα εξετάσετε μήπως ε, θα πρέπει να υπάρξουν πιο δεσμευτικά όρια. Να σας πω ευθύς ε, εξ αρχής το εξής. Συζητάω, ε, είμαι σε επαφή με τις εταιρείε, με τον κλάδο και ήδη διαμαρτύρονται αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν θα καταφέρουμε τίποτα αν δεν υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι. Γιατί λοιπόν εξακολουθούμε να επιμένουμε εφόσον ξέρουμε ότι θα, προκαλεί, θα σύγχυση. Έχουμε επιλέξει λοιπόν τέτοια κριτήρια για τα υγρά και βιοκαύσιμα. Γιατί δεν το επιλέγουμε αυτό και γιατί τα στέρεα βιομάζα. Μάλιστα λέει ο πρόεδρος, κανείς άλλος θέλει να θέσει ερωτήματα. Μάλιστα, να δώσω και πάλι το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει, αν θέλετε, μία ανακοίνωση ερμηνείας του νομικού κειμένου, το οποίο έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους δύο συνομοθέτες. Άρα δεν μπορείτε να αναμένετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση αυτή οτιδήποτε το οποίο θα φεύγει αν θέλετε από τα όρια του νομικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί αυτό τι σημαίνει. Χρειαζόμαστε κάτι το οποίο περιλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Άρα έχουμε περιορισμένο περιθώριο ελιγμών και τονίζω ότι αυτό το έργο διεξάγεται ως τώρα από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, όχι από τα κολέγια των Επιτροπών. Άρα μιλάμε για προκαταρτική ε, εργασία. Και γιατί καταρτήσαμε την ανακοίνωση αυτή, γιατί αποτελεί, αν θέλετε, μια κατευθυντήρια γραμμή για τα κρατημέλη, για τον κλάδο, για τους εμπλεκόμενους φορείς, για την εφαρμογή, τη μεταφορά της οδηγίας. Αλλά ασφαλώς δεν μπορεί να αλλάξει τις ε, καθεαυτές διατάξεις της ε, οδηγίας. Και η μόνη αρχή που μπορεί να κάνει τέτοια ερμηνεία και να προβεί σε τέτοια αλλαγή είναι το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τώρα, για τα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέσατε, σύμφωνα με τον κύριο Πρόντι και το σχόλιο που έκανε, ότι θα πρέπει να επιλύσουμε το θέμα αυτό των σχέσεων, αν θέλετε, της σύνδεσης, της ισορροπίας μεταξύ των ε, καλλιεργειών για τρόφιμα και για μη τρόφιμα. Αναφέρεται στην οδηγία ότι προβλέπεται ένα πόνους για την δεύτερη γενιά βιοκαυσίμων, όπως αναφέρεται, τα οποία παράγονται από την κυταρική αλυσίδα. Από τα υπολείμματα δηλαδή, της δασοκομείας και της ε, γεωργίας. Καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για την επιτάχυνση της εφαρμογής ε, των τεχνολογιών αυτών. για να μην επιβαρύνει περαιτέρω τις ε, καλλιέργειες τροφίμων. Άρα, Θεωρώ ότι υπάρχουν ήδη στην νομοθεσία κάποια νομικά κίνητρα για να ληφθούν υπόψη ε, οι ανησυχίες αυτές. Και επίσης υπάρχει και άλλο ένα κίνητρο. Αν οι καλλιέργειες βιοκαυσίμων, οι οποίες έχουν καλλιεργηθεί σε μολυσμένο έδαφος, αυτό, από ό,τι καταλαβαίνετε, απαντάει στα μελήματα που εκφράσατε. Τώρα, σχετικά με την ερμηνεία που δίνουμε στις φυτίες φοινικόδεντρων. Ακολουθούμε αυτά που αναφέρονται στο κείμενο. Συνεχώς δασωμένες περιοχές. Ε, δεν αναφέρεται η λέξη δάσος δηλαδή, όπως θα δείτε και στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές. Και γι' αυτό οι υπηρεσίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθούν να εξηγήσουν, να ερμηνεύσουν τον όρο αυτό. Αυτό που είπα και προηγουμένως είναι το εξής. Ανεξάρτητο αν πρόκειται για δασική περιοχή η φυτή αφηνικό το επίπεδο ε, αερίων ε, θερμοκηπίου που τύφεται ως προδιαγραφή δεν πληρείται κατά την μετατροπή φυτιών φυνικόδοντρων σε τέτοιες περιοχές. Άρα θεωρούμε ότι δεν θα πληρούνται έτσι οι όροι οι διατάξεις που προδιαγράφει η οδηγία. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι υπό εξέταση ακόμη από τι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιομάζα τώρα. Αντιλαμβανόμαστε και γνωρίζουμε την τοποθέτηση του κλάδου καθώς και τις ανησυχίες πολλών κρατών μελών. Ωστόσο, εξετάσαμε προσεκτικά το θέμα αυτό γιατί η κατάσταση ελαφρώς διαφέρει από τη βιομάζα, δηλαδή την υγρή. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη κυκλοφορία εισαγωγέ, εξαγωγές και εμπορικές ανταλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. γιατί η βιομάζα, σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές της βιομάζας, είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα τώρα, 5% περίπου. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της βιομάζας παράγεται στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους κοινωτικούς όρους. Θεωρούμε ότι αυτοί προστατεύουν επαρκώς την αεφορία της παραγωγής αυτής. Ως εκ τούτου, δεν θελήσαμε να επιβάλλουμε περιττό άχθος στους Ευρωπαίους παραγωγούς, που πολύ συχνά είναι πολύ μικροί, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά τέτοιες ε, απαιτήσει, αλλά παρακολουθούμε πολύ στενά την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. για να δούμε κατά πόσον υπάρχει ανάγκη περαιτέρω νομοθετικής ε, δράσης. Θεωρούμε λοιπόν ότι ήταν ε, μάλλον ε, συνετή και προσεκτική η προσέγγιση μας. Τώρα να δώσω τον λόγο στον συνάδελφο για να σας απαντήσει στα υπόλοιπα ερωτήματα. Thank you very much. Um, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον το οποίο δείχνεται στην αναλυτική εργασία και στη μοντελοποίηση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο το θέμα αυτό. Τι προσπαθεί λοιπόν να κάνει στην παρουσιαφάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να κατανοήσει καταρχάς την κλίμακα του φαινομένου Πρόκειται για μεγάλο, μικρό πρόβλημα. Όταν ε, το διαπιστώσουμε αυτό, μπορούμε να αποφανθούμε κατά πόσον χρειάζονται, αν χρειάζονται νομοθετικά μέτρα. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε να κάνουμε στην παρούσα φάση, με τις ε, ασκήσεις μοντελοποίησης αν θέλετε, είναι να κατανοήσουμε την έκταση, την κλίμακα του φαινομένου γίνονται διάφορες ε, ασκήσεις, αν θέλετε, στην παρούσα φάση. Καμία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη προκειμένου να μας ε, ε, δώσει επαρκή πορίσματα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπό έχει να διοργανώσει μια δημόσια διαβούλευση όταν θεωρήσει ότι έχει δημιουργηθεί βάσει της ανάλυσης η απαραίτητη επιστημονική βάση. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι η κατάλληλη στιγμή αυτή τώρα για να ξεκινήσουμε συζήτηση για το προς τα που οδεύουν και πώς διαμορφώνουν τα διάφορα μοντέλα. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο το θέμα, όπως σας είπα. Τα αποτελέσματα ως τώρα μας έχουν καταδείξει ότι υπάρχουν πολλές μεταβλητές, μικρότερες και μεγαλύτερες, και θεωρούμε ότι στην παρούσα φάση αυτό ε, προκαλεί μεγαλύτερη σύγχυση παρά διαλευκάνει το θέμα. Δεν θα ήθελα λοιπόν να επεκταθώ στο θέμα αυτό. Μπορώ να σας δώσω κάποια επιπλέον στοιχεία, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά τα δέντρα, να σας δώσω και κάποια αριθμητικά στοιχεία για το πόσες φυτίες χρησιμοποιούνται για βιοκαύσιμα επί του παρόντος. Μιλάμε για αριθμητικά στοιχεία τα οποία είναι ενδιαφέροντα, γιατί καταδεικνύουν ότι είναι πολύ περιορισμένος. Είναι περιορισμένο το τμήμα του φινικέλεου που χρησιμοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο για βιοκαύσιμα. Και συμφωνώ ότι υπάρχει μία ανησυχία για την επέκταση των φυτιών σε ό,τι αφορά τα τροπικά δάση, αλλά η πλειονότητα της αύξησης της συζήτηση για το φινικέλαιο δεν προέρχεται από τον τομέα της ενέργειας, προέρχεται από άλλους τομείς. Ε, αν θέλετε, έχω τα αριθμητικά στοιχεία, μπορώ να σας τα δώσω, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ίσως όχι τώρα. τώρα. Θέλει να προσθέσει κάτι ο κύριος Όαν από τη Γενική Διεύθυνση Κλιματικών Δράσεων. Όχι, ο κύριος Έκχαου τότε. Ευχαριστώ για τι απαντήσεις. Θα δώσω και εγώ μία μικρή, ένα μικρό σχόλιο. Γιατί κατάσταση σαφέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι απαντήσει τη ότι μιλάμε για ένα θέμα ορισμού στο φινικέλαιο. Αυτό είναι εν μέρη σημαντικό και στι πιο πολλέ περιπτώσει ε, δεν ισχύει. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ένα καλό ορισμό για το φινικέλαιο και ότι χρειάζεται σε κάποιες περιπτώσεις να έχουμε ένα καλό ορισμό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση και όλοι φυσικά αντιλαμβανόμαστε ότι χρησιμοποιείται για πολλούς άλλους σκοπούς το φινικέλαιο. Γι' αυτό όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί σε ό,τι αφορά τον ορισμό των φυτιών φοινικών Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μετακινείται ακόμα και ελαφριά αυτός ο ορισμός. Θα ήθελαμε λοιπόν να είναι πάρα πολύ αυστηρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τον ορισμό των φοιτιών αυτών για να μην περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση δάση. Για τις δημόσιες διαβουλεύσεις τώρα, νομίζω ότι καταδεικνύουν σαφές, σαφώς ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις αυτές. Όλα τα μοντέλα σε κάθε περίπτωση ωστόσο καταδεικνύουν ότι υπάρχει αντίκτυπος. Γι' αυτό λοιπόν ανυπομονώ να δω τι θα, ποια θα είναι τα πορίσματα των διαβουλεύσεων στο Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή με το κοινό. Ευχαριστώ πολύ. Um, Ευχαριστώ. Είχα μία ερώτηση στο προηγούμενο γύρο και δεν μου δόθηκε απάντηση. Το ερώτημά μου είναι κατά πόσο αποκλείεται ότι το φινικέλαιο που προέρχεται από μια φυτεία η οποία ήταν δάσος θα ενταχθεί στα κριτήρια βιωσιμότητας. Νομίζω το ερώτημα είναι απόλυτα σαφές. Η Κομισιόν. Θα θέλατε μία καταφατική αρνητική απάντηση με ένα ναι ή όχι. Αλλά όσοι είδατε το πρόγραμμα βιωσιμότητας γνωρίζετε ότι πρόκειται για μία περίπλοκη περίπτωση. Υπάρχουν τρία κριτήρια. Το κριτήριο της βιοπικιλότητας, δηλαδή ο, ορισμένες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βιοκαύσιμα. Άρα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν βιοκαύσιμα εκεί που ήταν τροπικά ε, δάση. Υπάρχει και το θέμα της, του υπολογισμού εκπομπών ε, αερίων θερμοκηπίου, όπου γίνεται ένας περίπλοκος ε, υπολογισμός και όλα εξαρτώνται από τη μεμονημένη περίπτωση για να δούμε κατά πόσο αυτό το κριτήριο ισχύει για τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Και το άλλο κριτήριο είναι κατά πόσο γίνεται αποθήκευση άνθρακα. Ε, για να δούμε κατά πόσο αφορά αυτές τις καλλιέργειες ή υγιές. Γι' αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω με ένα ναι ή όχι σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ότι επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται. Αλλά θα ήθελα να προσαφηνήσω κάτι στο οποίο αναφέρθηκα πριν ως προς την ενεργειακή χρήση και τις άλλες χρήσεις. Εδώ μιλάμε για, το κατά πόσο μπορούν να παραχθούν βιοκαύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς, με βάση δηλαδή τη στοχοθέτηση αυτή. Το φινικέλαιο με βάση τις περισσότερες ποσότητες δεν υπάρχουν κριτήρια βιωσιμότητας και αυτό θα πρέπει να έχετε κατά νου όταν συζητάμε παρεμφερή ζητήματα. Ωραία. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις ε, διεθνείς ε, εμπορικές συμφωνίες. Ε, Τόμας Άλμερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ έχουμε να γνωρίσουμε για την Επιτροπή Εξωτερικών Εμπορικών Σχέσεων όσον αφορά την εφαρμογή των ε, κοινωνικών ε, προτύπων και των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, μετά τις συνθήκες της Λισαβόνας όπου μπορούμε να, πρέπει να εγκρίνουμε εμπορικές συμφωνίες και έχουμε λοιπόν περισσότερο λέγει στο τομέα αυτό. Εγώ θεωρώ ότι μέτρα για την συμπερίληψη των κοινωνικών αυτών προτύπων και προτύπων της ε, ε των ζώων θα πρέπει να συμπεριληφθούν και θα ήθελα να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε κάτι τέτοιο στις εμπορικές ε, συμφωνίες. Χρειαζόμαστε και μία μέθοδο εποπτείας και θα ήθελα να σας πω ότι αν θέλουμε τώρα να έχουμε μία διεθνή εναρμόνιση των περιβαλλοντολογικών ε, προτύπων θα αποτύχουμε. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να επιδιώκουμε μια πλήρη εναρμόνιση. Αυτό ίσως μετά από 20 χρόνια θα μπορεί να γίνει. Επίσης χρειαζόμαστε νομίζω μια υπηρεσία διαιτησίας για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι και γενναιόδοροι όσον αφορά τις χώρες ε, του κατοφλίου και μέσα στα πλαίσια της οικονομικής ε, κρίσης θα πρέπει να προσπαθήσουμε μέσα στα πλαίσια διαπραγματεύσεων ΠΟΕ να έχουμε υπόψη μας ότι δεν πρέπει να προσπίζουμε κυρίως τα εμπορικά και οικονομικά συμφέροντα, αλλά και το θέμα της αηφορίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και άλλα παρόμοια κριτήρια. Θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι πιστεύουμε ότι τα κριτήρια αυτά δεν θα παρεμποδίζουν τις ελεύθερες διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να, όταν αποστέλουμε παρατηρητές ε, για τις συμφωνίες αυτές να έχουν πρόσβαση σε όλες τις συνεδριάσεις, να είναι πλήρως ενήμεροι. Αυτό το απαιτεί εκτός αυτού και η συνθήκη της Λισαβόνας. Είμαι ανοιχτός για κάποια πρόταση που μπορείτε να έχετε. Ευχαριστώ. Oh, uh, for the shadows, first Mr. Prodi. Ο κύριος Πρόντι καταρχήν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ούλμερ που έθιξε αυτό το ζήτημα ουσίας. Εγώ το συσχετίζω με το European Emission Trading System, δηλαδή το σύστημα ανταλλαγών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση να προβεί σε μία ανασύσταση αρμοδιοτήτων στον τομέα αυτό Ο ΠΟΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καθώς και η Παγκόσμια Τράπεζα είναι οργανισμοί που την χάνουν αυτόνομης διαχείρισης μεταξύ τους. Δεν μπορούμε όμως να μην λάβουμε υπόψη μία συντονισμένη διαχείριση διότι αν δούμε το θέμα της πειθαρχία των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν ε, ε, οργανισμοί οι οποίοι προβάλλουν κυρώσεις κατά μιας ορισμένης συμπεριφοράς, και αυτό αφορά ιδιαίτερα τον ΠΟΕ, διότι Δεν μπορεί να μην υπάρχει κάποια κύρωση, να μην υπάρχουν κυρώσεις σε σχέση με τα τέλιστα στα σύνορα για τις χώρες που δεν δεν επιμερίζονται μάλλον αυτές τις ευθύνες. Δεν μπορούν να μην δίνονται και κίνητρα. Κίνητρα καθαρά οικονομικά τα οποία να εγγυάται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή Παγκόσμια Τράπεζα. Άρα, έτσι θα πρέπει να τεθεί το ζήτημα και θα πρέπει να το κάνουμε με αυτή την ευκαιρία, διότι αυτό το σύστημα το διαχειριζόμαστε, θα πρέπει να το διαχειριστούμε συντονισμένα. Διαφορετικά δεν θα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε αυτήν την κατάσταση αλληλεξάρτησης που είναι απόλυτα σαφής ε, ως προς το θέμα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και ως προς το θέμα της ε, συμμεριζόμενης διαχείρισης των ε, εκπομπών αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να φτάσουμε σε μία συστημική συμμετοχή όλων των ε, διεθνών οργανισμών για να κατανείμουμε τις ευθύνες. Και θα πρέπει να προβάλλουμε ένα σύστημα παγκόσμιας διαχείρισης, διακυβέρνησης που να λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία. Ο κύριος Στάς. Ο κύριος Βαντάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Ούλμερ προέβαλε πολύ ενδιαφέρουσες ε, υποδείξεις. Δεν ξέρω πώς θα απαντήσει η Επιτροπή σε λίγο. Θα ήθελα να του ζητήσω ορισμένες αποσαφηνήσεις επίσης σε σχέση με το τέταρτο σημείο που ανέφερε, δηλαδή την εναρμόνιση των ε, προδιαγραφών υγείας και υγιεινής που δεν θα πρέπει να γίνει αποδεκτή. Τι σημαίνει, τι εννοεί μάλλον με αυτό. Εννοεί, μιλάει για τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τους ε, παγκόσμιους κανόνες στο έκτο σημείο των προτάσεών του μιλά για προτίμηση στις αναδιόμενες χώρες. Τι εννοεί και μιλάτε για τις άρτη βιομηχανιστήσεις χώρες χωρίς εξαίρεση. Επίσης είναι σαφές τι εννοούμε ακριβώς, ότι έχουμε έναν ενιαίο ορισμό για τις νεοεκβιομηχανιστήσεις χώρες. Στην ένατη υπόδειξη μιλά για την αποτίμηση των μέτρων και όπως λέει και στο τέλος θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή αυτών των κανόνων όχι μόνο δηλαδή ότι εφαρμόζονται, αλλά θα πρέπει να φτάσουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και κυρώσεις, αν δεν ακολουθεί κανείς τους κανόνες. Δεν είμαι σίγουρος ότι ακριβώς αυτό εννοεί ο εισήγητης. Είναι το θέμα ένα θέμα καθαρά διατύπωσης ή θα υπάρχουν ε, ρητές κυρώσεις για αυτούς που δεν θα εφαρμόζουν τους κανόνες. Ehm, Ευχαριστώ. Η κυρία Παρβάνοβα, η Σκιώδης, ε, δεν είναι παρούσα, γι' αυτό θα την εκπροσωπήσω εγώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, έκθεση του γενικά, η οποία μας βρίσκει σύμφωνους. Θα πρέπει να ξέρουμε γιατί υπάρχει ΠΟΕ. Καταρχήν θέλουμε περισσότερο εμπόριο, περισσότερη ευημερία, περισσότερη αηφορία. Αυτό σημαίνει καθαρό περιβάλλον πρωτίστως. Αυτό συμβαδίζει με τους άλλους στόχους του ΠΟΕ. Εμείς ως φιλελεύθεροι είμαστε πεπισμένοι ότι μια σωστή εμπορική πολιτική προστατεύει ακόμα περισσότερο το περιβάλλον. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο σε επίπεδο ΠΟΕ για να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Τα μέτρα αυτά όμως θα πρέπει να συμβαδίζουν με τους εμπορικούς κανόνες επί των οποίων συμφωνούμε όλοι. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή να καταστήσει σαφές το ΠΟΕ ότι οι περιβαλλοντικές, ε, η περιβαλλοντική αυτή συλλογιστική είναι θεμητή και θα πρέπει να διέπει και τις ε, διεθνείς συμφωνίες εμπορίου. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή, να ζητήσω από την Επιτροπή να σχολιάσει. Ο κύριος ε, Σάντσες ε, έχει το λόγο από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή, ευχαριστώ. Λάβαμε υπόψη την πρόταση γνωμοδότησης και συμφωνούμε με τους απότερους στόχους και την κατεύθυνση του όλου εγχειρήματος και εμείς προωθούμε μια πολιτική που λαμβάνει υπόψη την ε, περιβαλλοντική αυτή πτυχή για να προωθήσουμε την ε, προστασία του περιβάλλοντος κατά τις ε, διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες. Και θα το λάβετε κι εσείς αυτό όταν ασχοληθείτε με τις διμερείς ή πολυμερείς αυτές συμφωνίες. Αυτός είναι κοινός στόχος από την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Τώρα, σε σχέση με τα συγκεκριμένα θέματα στην γνωμοδότηση, έχουμε ορισμένα σχόλια. Δεν θα μακρηγορήσω. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι η Επιτροπή έχει ορισμένα ερωτήματα, όπως ε, στην κατεύθυνση του κ. Παντόλεν, Δηλαδή, όταν μιλάμε για εναρμόνιση περιβαλλοντικών κανόνων και κανόνων υγιεινής, μιλάμε σε παγκόσμιο ε, επίπεδο και όχι σε ευρωπαϊκό. Γιατί εμείς έτσι κι αλλιώς εναρμονίζουμε ό,τι μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως προς τις ε, προτιμήσεις σε χώρες κατοφλίου, Εάν λάβουμε υπόψη το γενικό σύστημα εμπορικών προτιμήσεων, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τη συζήτηση που γίνεται σε σχέση με την αναθεώρηση του ΓΚΑΤ και εσείς θα ασχοληθείτε με αυτό το ζήτημα λίγο αργότερα. Θα χρειαστούν ε, μακροσκελής διαβουλεύσεις, άρα πρωταρχικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό το ζήτημα ίσως θα, το, θα μπορούσε να ειδωθεί στα ευρύτερα αυτά πλαίσια των εμπορικών προτιμήσεων. θεωρούμε ότι και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό θα είναι το θέμα μιας ειδική διαπραγμάτευσης μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για να λάβουμε υπόψη τα νέα στοιχεία της συνθήκης της Λισαβόνας, από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Άρα η συνθήκη θα ορίσει την φύση της συμμετοχής, το βαθμό συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τις συναντήσεις και διαπραγματεύσεις. Τέλος, The World Organization has a competence Ο ΠΟΕ έχει βασικό ρόλο ως πραγματογνώμονας γιατί πρόκειται για εμπορικούς κανόνες στο κάτω-κάτω. Θα πρέπει να ελέγχει τη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις στα πλαίσια και των διμερών συμφωνιών, ως προς τις πολυμερείς αυτό καθίσταται πιο δύσκολο. Ως προς τα σώματα διαιτησίας και εφαρμογής υπάρχουν ειδικέ διαδικασίες διαιτησίας για να δούμε κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με περιβαλλοντικά κριτήρια στις ε, διμερείς συμφωνίες και η διαιτησία είναι δεσμευτική. Άπαξ και έχει ξεκινήσει, οι χώρες θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία. Βεβαίω δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα συμμορφωθούν οι χώρες με ένα ε, διεθνές σώμα διαιτησίας σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία και ε, την ιατρική θεώρηση του θέματος. Αυτό κινείται λίγο πέραν του περιβαλλοντικού στις εμπορικές συμφωνίες. Βεβαίως υπάρχει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ περιβάλλοντος και ανθρώπινης υγείας, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις υψηλές προδιαγραφές περί ανθρώπινης υγείας και εκτινιατρικής υγείας θα εφαρμόζει αυτά τα κριτήρια. Και ξέρουμε ότι στην περίπτωση εισαγωγών, οι εισαγωγές θα πρέπει να συμμορφούνται με τα δικά μας κριτήρια περί ανθρώπινης υγείας και θεμάτων υγιεινής. Το περιβαλλοντικό είναι λίγο διαφορετικό, αλλά η Επιτροπή το περιλαμβάνει στις εμπορικές συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Ευχαριστώ κύριε Πατέρα Σέντρες. Το λόγο έχει ο Τόμας Ούλμερ για να ολοκληρώσουμε. Ναι, ευχαριστώ και πάλι Πρόεδρε. Θα συμπεριλάβω και κάποιες τροπολογίες για να είναι πιο σαφές ε, το θέμα. Δεν έχουμε βέβαια πολλές λεπτότητες να πούμε πολλά σε μια γνωμοδότηση. Σημείο 4 προφανώ είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για διεθνή πρότυπα. Το σημείο 6 με αυτό το σύστημα πρέπει να διατυπωθεί. Στο σημείο 9 όσον αφορά τα σκερώσεις εγώ δεν τις έχω απαριθμίσει. Θα το κάνω. Μου φαίνεται ότι είναι σωστό να μην έχουμε μονάχα μια εποπτεία, αλλά να έχουμε και ένα κατάλογο για να μπορούμε να τονίσουμε ε, καλύτερα αυτό που εννοούμε. Λόγω του συντόμου του κειμένου δεν έχω αναφέρει τίποτα για το εμπόριο των εκπομπών αερίου. Θα ήταν καλό κάπου να μπορέσουμε να το αναφέρουμε και αυτό μέσα στα πλαίσια αυτή της έκθεση πρωτοβουλία. Και με χαρά θα περιμένω τις ε, τροπολογίες σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Η προθυμία για την υποβολή των απολογιών είναι 18 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι και η ψηφοφορία στις 27 Μαρτίου στην Επιτροπή μας. Α, όχι, Απριλίου. Απριλίου. Ναι. 27 Απριλίου έκανα λάθος. Περνάμε τώρα στο σημείο 8 της υπηρεσίας διάταξης. Παροχή πληροφοριών για το τρόφιμο στους καταναλωτές. Ένα θέμα που έχουμε συζητήσει πριστάκες και αύριο θα περάσουμε και στην ψηφοφορία. Η συζήτηση σήμερα έχει σαν ε, νόημα να δούμε ποιε είναι οι συμβασικέ τροπολογίε που υπάρχουν. Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Μία ώρα έχουμε χρόνο γι' αυτό. Θα έλεγα να μην μιλήσει κανένα πάνω από πέντε λεπτά. Η συγγήτρια κυρία Σόμερ είναι απασχολημένη σε συζήτηση με τη γραμματεία. όπου ο κύριος Ράιερ προετοίμασε τον κατάλογο της ψηφορίας το Σαββατοκύριακα. 800 τροπολογίες υπήρχαν. Σας ευχαριστώ ήδη τώρα και ελπίζω να, μπορέσουμε να ψηφίσουμε πολύ καλά αύριο. Λοιπόν, του των. Η κυρία Σόμερ θα μπορούσαμε να μας παρουσιάσει τι γίνεται. Πέντε λεπτά, οι πέντε λεπτά και μετά βλέπουμε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πράγματι, όλο το Σαββατογικό δουλέψαμε και θα ήθελα να ευχαριστήσω την γραμματεία που μας έδωσε τη δυνατότητα αυτό. Και γι' αυτό βέβαια ο κατάλογος ψηφοφορίας μόλις τώρα προετοιμάστηκε. Ε, αυτό το ξέρουμε βέβαια και από άλλες τροπολογίες και φακέλους πολύ ογκώδης. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ μην ξεχνάτε ποτέ και δεν το βλέπω σε διάφορες τροπολογίες ότι αυτή η πρόταση κανονισμού βέβαια είναι προς όφελος του καταναλωτή, ούτως ώστε ο καταναλωτής να έχει πιο ευανάγνωστε και ευνόητε πληροφορίε στα τρόφιμα Από την άλλη μεριά, βέβαια, αυτή η πρόταση θα πρέπει να καλύψει και τις ανάγκες ε, ε, της άλλης πλευράς, δηλαδή της εσωτερικής αγοράς. Ε, ανάλογα βέβαια θα δούμε κατά πόσο θα υπερψηφίσουμε τις τροπολογίες ή όχι. Τι γίνεται τώρα, υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις στο φάκελο αυτό έχουμε προσεγγίσει αρκετά. Μπορούμε και ορισμένες να ε, είναι πιο ευανάγνωσες. Αν δείτε τα τρία χιλιοστά παραδείγματος χάρη προτείνει η Κομισιόν για το μέγεθος των γραμμάτων και επίσης το σημείο της ε, παραπληροφόρησης στο άρθρο 7. Κανένας δεν θέλει βέβαια να παραπληροφορηθεί ο κατανοτής και εκεί είμαστε πολύ πλησίοι με τις ιδέες μας. Σε άλλα σημεία όμως δεν συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν διάφορες θέσει παραδείγματο χάρη για την σήμανση τη προέλευση. Ορισμένοι λένε να λέγεται προέλευση ε, για το βόλιο κρέα που έχει διακανοστεί μέχρι όλα τα άλλες τη πρώτη μέχρι τα χαρακτηριστικά υλικά στα επεξεργασμένα προϊόντα και ούτω καθεξής. Εγώ δεν έχω ένα πρόβλημα με την σήμανση προέλευσης, αλλά ξέρω ότι αυτό δεν είναι προς όφελος του κανονιστή από τη ΦΕΝΤΗ γιατί έχει γίνει μια έρευνα από την Βρετανική FSA, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των κατανοτών ενδιαφέρεται για την προέλευση των τροφίμων τους. όλα αυτά θέλω να τους δώσω τις πληροφορίες αλλά θα ήθελα να συμφωνήσουμε να κάνουμε καταρχήν μία εκτίμηση από την Κομισιόν κατά πόσο αυτό είναι δυνατό και ποιες θα είναι οι ενδεχόμενες δυσκολίες όσον αφορά τα, τις πρώτες ύλες, αλλά και ίσως και κάποια συγκεκριμένα συστατικά. Δεν ήθελα να με υποστηρίξετε σε αυτή την ιδέα. Πρώτα να κάνουμε μία εκτίμηση των συνεπιών. Κατά πόσο αυτό μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Υπάρχουν διαφορετικέ απόψεις όσον αφορά το θέμα των εθνικών συστημάτων σύμμαξης. Η Κομισιόν προτείνει τα κράτη-μέλη να είναι ελεύθερα να αναπτύξουν μη υποχρεωτικά εθνικά ε, συστήματα σήμανσης. Εγώ φοβούμαι ότι αν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι ε, εις βάρος της εσωτερικής αγοράς, γιατί αλλιώς θα καταλήξουμε να έχουμε 27 συστήματα σήμανσης που δεν θα είναι υποχρεωτικά νομικά δεσμευτικά, αλλά βέβαια de facto στα κράτη-μέλη θα είναι δεσμευτικά. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακλώσω να μην το επιτρέψουν αυτό και το είπανε και αυτές οι δύο συνοδευτικέ επιτροπέ, ΙΜΚΟ και Άκρη, που απέριψαν για αυτό το λόγο αυτά τα λεγόμενα εθνικά συστήματα. Η δε, δεύτερη εξαίρεση από τον κανονισμό. Εγώ θα ήθελα τα μη ε, συσκευασμένα προϊόντα, τα ψωμάκια στον στο φούρνο ή το φρέσκο κρέας στο χασάπι να εξαιρεθούν από το κανονισμό αυτό. Δηλαδή, οι... εκείνοι που προσφέρουν τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να πληρούν τους όρους της οδηγίας. Αυτό που θα μπορούσε να υπάρχει είναι πληροφορία για αλλεργογόνα, αλλά όποιος έχει διαβάσει τις ε, τροπολογίες ε, θα δει ότι εγώ προτείνω κάτι διαφορετικό Στη συζήτηση παραδείγματος κάνουμε με το προσωπικό, με ανακοίνωση μέσα στο κατάστημα ή κάπως διαφορετικά. Βέβαια στα μη προσυσκευασμένα προϊόντα συμπεριλαμβάνεται και το φαγητό στα εστιατόρια. Εάν δεν τα εξαιρέσουμε θα τρώμε παντού τα ίδια, δηλαδή θα βγαίνουν τα φαγητά από, το... από την κατάρτιση, θα μπαίνουν στα μικροκύματα και θα τρώμε παντού τα ίδια πράγματα και δεν θέλουμε αυτό. Μετά το θέμα των ε, ε, το ότι δεν θέλουμε να εξαφανιστούν οι περιφερειακές, ε, ε, τα περιφερειακά τρόφιμα, σπεσιαλιτέ αν θέλετε, από την αγορά. Βέβαια δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε. Μην ξεχνάμε στην εορτή της μητέρας, ας πούμε, ε, άμα η μαμά μου το πρώτο που θα κοιτάξει στα σοκολαράκια που τα σχαρίσω είναι τι περιέχουν τα σοκολατάκια αυτά, δεν θα ήταν και πάρα πολύ ωραίο. Περαιτέρω. Προτείνω να μην υπάρχει αυτό που είχαμε στην λεγόμενη health claim ε, κανονισμό. γιατί μέχρι στιγμής αυτά τα στοιχεία δεν έχουν συμπεριληφθεί ε, και η Κομισιόν ένα χρόνο μετά που υπάρχει αυτός ο, ο, ο κανονισμός έπρεπε να είχε δημοσιεύσει, δημοσιεύσει αυτά τα προφίλ. Φαίνεται όμως ότι δεν έγινε γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί ε, στην πράξη. Τελειώνω Πρόεδρε. Η Κομισιόν σε μία επερώτηση απάντησε ότι θα ήθελε να παρεμποδίσει τις δηλώσεις αυτές ε, σε κίτρινο, πράσινο, κόκκινο. Θα είχε μόνο πράσινο στην περίπτωση αυτή. Παρακαλώ να υποστηρίσετε όσον αφορά αυτή η δεν εξαφανιστεί. Όσον αφορά την υποχρεωτική αυτή σήμαση με τα τρία χρώματα αυτά κόκκινα πορτοκαλί και πράσινο. Αυτό δεν επιτρέπεται να υπάρχει γιατί θα ε, παραπληροφορήσει έτσι τον, ε, τον καταναλωτή και δεν θα τον ωφελήσει καθόλου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σόμερ. Περνάμε στους κοιόδες ηγητές. Κρίνης Φίλμετ. Είχαμε συζητήσεις για την σήμανση προϊόντων και δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά τα επιχειρήματα, γιατί τα έχουμε αναφέρει πολύ. Αλλά πολλοί εξέφρασαν ανησυχίες και νομίζω θα πρέπει να έχουμε ορισμένες ενοποιημένες τροπολογίες. Η πρώτη αφορά τη χώρα προέλευσης και στάλει αυτή η τροπολογία είναι υπαριθμόν 2 είναι πιο πρακτική προσέγγιση από ορισμένε άλλες τοπολογίε, γιατί δεσμευτικά θα μιλάμε για χώρα προέλευση, για τα νοπά οποροκυπευτικά, όλων των ειδών τα κρέατα, για το βόλιο κρέας και τα ψάρια είναι δεσμευτικό, ε, θα είναι και για τα πουλερικά και όσοι παρασκευαστές λένε ότι είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν ε, πολυπληθείς πηγές, μπορούν να μιλάνε για μη ορισμένη, μη ορισμένη εκ των προτέρων προέλευση. Επίσης, ως προς το, τις υποχρεωτικές πληροφορίες διατροφής, αυτό δεν θα ισχύσει για προϊόντα όπως τον άρτο, το γάλα, τους χυμούς φρούτων, αλλά μόνο για τα μεταποιημένα προϊόντα όπως τα έτοιμα γεύματα. Αυτή είναι η τελική τροπολογία και νομίζω ότι είναι καλύτερος τρόπος, δηλαδή λαζάνια κλπ. Έτοιμα γεύματα. Ως προς την εννέα, ζήτησα από την Επιτροπή να μας δώσει κατευθυντήριες γραμμές για ε, μερίδες τι εννοούμε με μερίδες, αυτό να μας το ορίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι ε, φορείς και ιδιαίτερα σε σχέση με την ε, ε, θερμιδική αξία των προϊόντων αυτών. Δηλαδή θα ορίσουμε θερμιδική αξία με βάση τα δεδομένα της ΕΦΣΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων. Εάν δεν υποστηρίξετε τις υποχρεωτικές αυτές πληροφορίες, μην ξεχνάτε ότι θα συνεχίσουν τα εθνικά προγράμματα. Άρα δεν θα πρέπει να επιτρέψετε σε ορισμένα κράτη-μέλη να μην δίνουν αυτές πληροφορίες. Τέλος, οι καταναλωτές θέλουν πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης, για τη θερμιδική αξία την ε, διατροφική αξία και θεωρούμε ότι είναι μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για παχυσαρκία, για καρδιακές ε, παθήσεις, ε, διαβήτη και ούτω καθεξής. Εφόσον θέλουμε να αντιμετωπίσουμε θέματα υγείας, τότε θα πρέπει να έχουμε αυτές τις πληροφορίες που θέλουν και οι καταναλωτές για να προβούν σε επιλογές στο τομέα της υγείας και υγιεινής. Πολλά λόμπι έχουν ε, δράσει και οι ενός καταναλωτών δεν έχουν τα ίδια μέσα. Όταν αποφασίσετε για αυτές τις πληροφορίες σκεφτείτε προσωπικά, ε, προσεκτικά. Ε, θέλετε να ακούσετε τα λόμπι του βιομηχανικού τομέα ή θέλετε να προωθήσετε τις ε, πληροφορίες που θέλουν οι καταναλωτές και οι φορείς υγείας και υγιεινής. Διότι αυτά τα στοιχεία είναι χρήσιμα για τον καταναλωτή για να προβεί σε σωστές επιλογές. Δεν πρέπει να, ακούμε, να εισακούονται πάντα τα λόμπι του βιομηχανικού τομέα. Perfect in time. Danke, Klenis. Ακριβώς ήρθε το χρόνο. Σε ευχαριστώ, Κλένης. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het niet eh, heel lang... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν πρόκειται να μακρηγορήσω, γιατί το έχουμε συζητήσει πολλά και στο θέμα αυτό. Και ένα από τα στοιχεία που μου έκανε εντύπωση τους προηγούμενους μήνες είναι το εξή. Οι θέσεις δεν έχουν τροποποιηθεί τους τελευταίους μήνες. Δεν πρόκειται να κάνουμε επαναλήψεις όμως. Φοβάμαι, ή μάλλον το πω αλλιώς, είναι θετικό το γεγονός ότι σε κάποια θέματα έχουμε κάποιες consolidated, όπως τις λέμε, επιμένες τροπολογίες. Αυτό θα απλοποιήσει και θα επιταχύνει τη διαδικασία, ωστόσο δεν σημαίνει αυτό ότι προσεγγίσαμε κιόλα ε, ο ένα τον άλλον σε ό,τι αφορά τι απόψει μα και είμαι πεπισμένο ότι η πραγματική δουλειά θα ξεκινήσει ουσιαστικά μετά την αυριανή ψηφοφορία. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν μετά την ψηφοφορία ίσως να καταφέρουμε να συνάψουμε πραγματικούς συμβιβασμού. Μίλησα και με τον κλάδο αλλά και με τις ενώσεις καταναλωτών και ρώτησα κατά πόσον θα ήταν διατεθειμένοι να κάτσουν και να το συζητήσουν το θέμα αυτό μεταξύ τους. Γιατί αν εμείς δεν μπορέσουμε να υπερβούμε, αν θέλετε, τις ε, παροχημένες ε, εν μέρη θέσεις μα. Ε, ίσως θα μπορούσαν να μα βοηθήσουν αυτοί. Θα έδινε μια ενδιαφέρουσα τέτοια προοπτική στην ευρωπαϊκή πολιτική. Επαναλαμβάνω ότι αύριο θεωρώ ότι θα πρέπει να κάτσουμε να ψηφίσουμε αύριο τι πιο πολλέ ε, ψηφοφορίε, αλλά μετά ουσιαστικά θα ξεκινήσει η δουλειά της συμβιβασμού μεταξύ μα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Άρα δηλαδή από αύριο θα ξεκινήσει η πραγματική δουλειά, λέει ο Πρόεδρος. Θα συνεχιστεί το κεφάλαιο αυτό από τις άλλες ομάδες. Δεν έχουμε τους σκιώδεις εισηγητές, αλλά μπορεί να ζητήσει το λόγο όποιο θέλει. Αν σωστά κατάλαβα, υπάρχουν κάποιες προσεγγίσεις, συμφωνίες σε ό,τι αφορά τα θέματα αναγνωσιμότητας και της αποφυγής παραπλάνησης του καταναλωτή. Μόνο για αυτά δεν είναι και πάρα πολλά. Για τα υπόλοιπα δεν φαίνεται να δεν προδιαγράφονται καλά τα πράγματα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι έχει η κατάσταση. Η κυρία Χίμπνερ, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα αυτό και αυτό το μαρτυράει άλλωστε και ο αριθμός των τροπολογιών, πάνω από 800. Και μάλιστα το θέμα αυτό αφορά όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Εξαρτάται από το θέμα αυτό οι πληροφορίες που θα, λαμβάνει, θα λαμβάνουν όλες οι όλοι οι καταναλωτές. Αυτό δεν μπορεί να ξεπερνάει το ίδιο το μήνυμα. Όλα τα θέματα που ακούσαμε είναι λογικά και οι πιο πολλές τραπολογίες είναι λογικές, αλλά η 162 θα πρέπει να εξαφανιστεί, που μιλάει για τα θρεπτικά προφίλ. Και αν θέλετε, κάνει τις πληροφορίες που δίνονται υπερβολικές. Και προκαλούν και σύγχυση γιατί αυτό θα προκαλούσε διακριτική μεταχείριση κάποιων τροφίμων, το οποίο φυσικά είναι νοησία. Δεν νομίζω ότι σε ένα κανονισμό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί πραγματικά ένα τέτοιο άρθρο. Δεν έχει να κάνει αυτό τίποτα με οποιοδήποτε λόμπι κατασκευαστών παραγωγών. Δεν νομίζω ότι κάποιο λόμπι έχει συμφέρον να εισαχθεί αυτή η διατύπωση υπογείως. Το πρόβλημα όμως είναι ότι υπάρχουν κάποια κάποιες φράσεις, κάποιες διατυπώσεις αναφορικά με τις πληροφορίες και ασφαλώς ως καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουμε και να ενημερωνόμαστε για την θρεπτική αξία. Έχουμε το συντελεστή της ημερήσιας συνιστόμενης ποσότητας, το GDA και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί επαρκής, ε, επαρκής επίπεδο πληροφοριών όχι μόνο για τον καταναλωτή, αλλά και για τους ε, ειδικού θέματα διατροφής. Αν θέλουμε λοιπόν κάτι να αλλάξει, να τονίσουμε θέματα εκπαίδευσης. Η γενική διατροφή δεν ε, σημαίνει ότι θα δώσουμε όλες τις πληροφορίες πάνω σε ένα πακέτο. Δεν είναι δηλαδή, αν θέλετε, το κακό απαραίτητα η ζάχαρη ή το αλάτι. Θα πρέπει με καλύτερο τρόπο όμως να διοργανώσουμε τη διατροφή μας. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να αφαιρεθεί η 162 η τροπολογία. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος, ε, τρία λεπτά για τους ομιλητές. Λίζα, έχεις το λόγο. Ο κύριος Λίζα, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους ε, σκιώτες Ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο το έργο αυτό τα τελευταία χρόνια και τις τελευταίες ημέρες ε, ιδιαίτερα. Δύο πράγματα να τονίσω. Καταρχάς, ανεξάρτητα από το τι θα αποφασιστεί αύριο, τι θα αποφασιστεί στο τέλος της διαδικασίας αυτής, ο καταναλωτής θα λαμβάνει για τα τρόφιμα πιο πολλές πληροφορίες από ό,τι ως τώρα. Γιατί ως τώρα είχαμε κάποια θελοντικά συστήματα τα οποία είχαν εφαρμοστεί από κάποιες επιχειρήσεις εν μέρη με υποστήριξη άλλων ενώσεων, αλλά δεν υπήρχαν κοινοτικέ προδιαγραφές, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την αναφορά τη θερμητική αξία στην μπροστά πλευρά. Αυτό θα ακολουθήσει από το νομοθέτημα αυτό. Άρα σε κάθε περίπτωση θα είναι βελτιωμένε οι πληροφορίε που θα λαμβάνει Το δεύτερο, το οποίο ανέφερε η Ρενάντα Ζόμερ, να τονίσω επισταμένα, ότι πάρα πολύ συχνά μεγάλες ε, φίρμες, η Nestlé, οι Φεραίρο διακατέχουν τις ε, σκέψεις μας όταν συζητάμε, αλλά αυτά πλήττουν και εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά θα πρέπει να είναι εφικτά Σας παρακαλώ λοιπόν ως προς αυτά τα θέματα ιδιαίτερως να υποστηρίξετε την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος, η Κρίστα Κλάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν βρισκόμαστε στην αρχή της συζήτησης, ε, βρισκόμαστε εν το μέσο της συζήτησης. Ελπίζω αύριο να διαγραφεί και μια γραμμή, να μην ψηφίσουμε απλά αυθαίρετα και όπως είπε και ο κύριος Λίζα θα ακολουθήσει ένα φατικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τι πιστεύει ο καθένας, το γνωρίζουμε. Δύο τροπολογίες μας έκαναν εντύπωση σε ό,τι αφορά την επεξεργασία επιφάνειας οποροκυπευτικών, σε ό,τι αφορά τα φυτοφάρμακα και τα φυτοκτόνα, τα βιοκτόνα. Είναι πολύ σαφείς και αυστηροί οι κανονισμοί μας σχετικά με το τι επιτρέπεται ή όχι. Τώρα μία ετικέτα με την επεξεργασία της επιφάνειας δεν βλέπω τι προσφέρει στον καταναλωτή. Θα έπρεπε λοιπόν να αφαιρεθεί αυτή η αναφορά. Να τηρήσουμε λοιπόν τη γραμμή αυτή, ότι είμαστε αυστηροί ότι θέλουμε να διαβιβάζουμε τις σημαντικές πληροφορίες, όχι να παραπλανούμε τον καταναλωτή. Να τον ενημερώνουμε σωστά. Γιατί φυσικά αυτές οι επεξεργασίες ε, σκοπό έχουν να προστατεύσουν το φυτό, να καταπολεμήσουν τις μικροτοξίνες που φυσικά είναι αρνητικές για την υγεία. Άρα να μην ε, πλατιάζουμε στην ετικέτα, γιατί είναι και περιορισμένο ο χώρος που χρειάζεται. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται τέτοια αναφορά, λοιπόν, για την ε, επεξεργασία. Και μιλάμε για τις τροπολογίες 71 και 258. Ευχαριστώ, κύριος Σνέλχαρτ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορούμε να επενέσουμε την εισηγήτρια πολύ επιμελώς ε, εργάστηκε και υπάρχει στο, στην έκθεσή της μία ενιαία γραμμή. Η Ευρώπη αύριο θα κοιτάξει προς την Επιτροπή μας και έχουμε συγκεκριμένη ευθύνη στην οποία θα πρέπει να επεξέλθουμε. Θα πρέπει λοιπόν να τη δικαιώσουμε την ε, ευθύνη αυτή. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να, να επιβάλλουμε προβολικές απαιτήσεις στο Συμβούλιο. Δεν μιλάμε για δόγματα. Σας απευθύνω έκκληση. Δεν μιλάμε για ιδεολογίες. Μιλάμε για απλές και σαφείς πληροφορίες προς τον καταναλωτή, προκειμένου να επηρεάσουμε κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα, αν και αμφιβάλλω αν αυτό μπορεί να γίνει με επισήμανση. Για την επισήμανση νομίζω ότι προάγουμε και φοβάμαι ότι προάγουμε τον προστατευτισμό και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να καταστήσουμε υποχρεωτική αυτή την αναφορά προέλευση. Θεωρώ ότι δεν είναι κατάλληλη αυτή η επισήμανση και το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά θέματα υγιεινής τροφίμων. Τα μεγάλα προβλήματα δεν ε, παρουσιάζονται στα μεγάλα, στις μεγάλες εταιρείε, αλλά στις μικρές επιχειρήσεις, γιατί οι μικρές επιχειρήσεις απαρτίζουν ουσιαστικά, αν θέλετε, τη ραχοκοκαλιά της Ευρώπης και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε λοιπόν προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να μην τα συμπεριλάβουμε τα θέματα αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, επισήμανση του κρέατος. Ξέρω φυσικά ότι την χάνει κατάχρησης αυτή η επισήμανση, αλλά να μην προσπαθήσουμε να προβούμε σε περιττές ε, σε περιττούς ελέγχους. Θα πρέπει νομίζω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κοιτάξουμε και να το αφήσουμε αυτό το έργο στους ε, τοπικούς φορείς. Για ποιες τροπολογίες μιλάτε, λέει ο Πρόεδρος. 177. Μάλιστα. Η κυρία Πιλάρα Γιούζο. Το πρώτο είναι να ευχαριστήσω την κυρία Σόμερ για την ε, εργασία της και για τις κατευθυντήριες γραμμές που μας ε, δίνει. Συμφωνώ απόλυτα με τις προδιαγραφές αυτές. Θα ήθελα να διευκνήσω τα εξής. Τα κεφάλαια 6 και 7, εθνικά στοιχεία και εκτιμήσεις, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να γίνει εναρμόνιση. Εάν θέλουμε να γίνει μία αποσάφηση, τότε θα πρέπει να πάμε στην εναρμονημένη ε, ονοματολογία, τουλάχιστον ως προς αυτό το θέμα της ε, σήμανσης. Ως προς τη σήμανση, νομίζω ότι το άρθρο 16 της οδηγίας 2013 έχει εφαρμοστεί χωρίς ε, πρόβλημα και θεωρούμε ότι είναι επαρκές. Αυτό αφορά και την Κομισιόν και το Συμβούλιο, γι' αυτό θα πρέπει να το αφήσουμε ως έχει. Σε σχέση με τη σήμανση των αλκοολούχων ποτών και των ανθρακούχων αλκοολούχων, νομίζω ότι θα πρέπει να τα αφήσουμε κατά μέρος. Νομίζω ότι η έγκριση της τροπολογίας από την Επιτροπή ΙΝΚΟ ε, που αφορά τα συστατικά στοιχεία αλλά όχι τη διατροφική αξία είναι σωστό. Στον ε, τομέα το, της αγροτικής βιομηχανίας θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις ΜΜΕ έτσι ώστε να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικές. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Η Άνια Βαϊσκεύερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ καταρχήν να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια γιατί υπέβαλε μια πάρα πολύ καλή έκθεση και νομίζω ότι μας παρουσίασε και μια πολύ καλή γραμμή αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι αύριο θα πρέπει να υιοθετήσουμε κάτι που θα είναι καλό για τους καταναλωτές, γιατί αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε έναν ενήλικο καταναλωτή. Και παραδείγματο χάρη να ζητήσουμε να αναφέρουμε τις ε, θρεπτικές, ε, τα στοιχεία για τις θρεπτικές ουσίες ε, δεσμευτικά θερμίδες, ε, λίπη, πρωτεΐνες κλπ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους καταναλωτέ, και πρέπει να επιμείνουμε γιατί έτσι θα μπορέσει ο καταναλωτή να αποφασίζει εν γνώση του τι αγοράζει και να είναι πια ένας ενηλικιωμένος καταναλωτής όσον αφορά το θέραμα της αναγνωσιμότητας τις διάφορες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί από εμά και συζητηθεί είναι καλές λύσεις Στι συμβαστικέ τροπολογίε επίση είναι πολύ καλά. Όσον αφορά τι εξαιρέσει, θα ήθελα να τονίσω αυτό που είπαν οι συνάδελφοι προηγουμένω, ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια δυνατότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό έχουμε τις εξαιρέσεις για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα. Και τώρα θα ήθελα να στραφώ σε κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ καλά. Είναι η καλύτερη σήμαση των απομιμήσεων τροφίμων. Γιατί στην Επιτροπή ε, προστασία των καταναλωτών και στην Επιτροπή Άγκρη, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα θέμα για το οποίο μπορούμε να ευθυγραμμιστούμε. Όλες οι πολιτικές ομάδες έχουν συμφωνήσει με τις σχετικές τροπολογίες, όπως και η κυρία Σόμερ συμφώνησε. Υπήρχε ομόφωνη ψηφορία. Εγώ αναφέρομαι εδώ στην τροπολογία 68 της συγγήτριας με καλύτερη σήμαση από την εμφανή η 261 επίσης, όπου ορίζουμε τι είναι μια απομίμηση, η 271 που συμπεριλαμβάνεται στη συμβαστική, όπου λέμε ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει παραπληροφόρηση με τις εικόνες και 577 επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική προς την αυτή και υιοθετήθηκε ομόφωνα από την ΕΜΚΟ. Ε, αυτό είναι ένα θέμα όπου θέλουμε ομόφωνα να δώσουμε ένα μήνυμα ως κοινοβούλιο, γιατί ε, θα πρέπει να πετύχουμε και ομοφωνία στο Συμβούλιο αυτή τη στιγμή η Γερμανία, η Αυστρία και ίσως και η Ιταλία είναι υπέρ του θέματος αυτού. Αλλά θέλω να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες να ε, ευθυγραμμιστούν γιατί λέμε ότι δεν επιτρέπεται να παραπληροφορείτε, να απατείτε αν θέλετε ο καταναλωτής. Το είπε και ο Επίτροπος αυτό, παραδείγματο χάρη, όταν έχουμε ε, απομηνήσεις ε, τυριού ή ζαμπών και θα χαιρόμουν πάρα πολύ να με υποστηρίξουν εδώ οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής. Ρουσπέτερλε. Hvala Καλησπέρα, gospod predsednik. Jaz sem vesel ambicije poročevalke, da ne Χαίρομαι, διότι η συγγήτρια δεν θέλει να αναφερθεί μόνο σε καλές προθέσεις και να μην βρεθεί σε ακόμα δυσκολότερη θέση ο εισηγητής από αυτή που ήδη είναι. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε την αρχή της αναλογικότητας και χαίρομαι διότι δεν θέλετε να επαυξηθεί η γραφειοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Λαμβάνουμε υπόψη τις μικρομεσές, τους ε, μικρούς ε, παρασκευαστές ε, γευμάτων. Δεν θέλω να επιδεινώσω τη θέση της εισηγήτριας, αλλά ως μελισσοκόμος Προσπάθησα να βρω το δρόμο μου μέσα σε αυτή την, ε, ε, μεγάλη, τη μεγάλη επιφάνεια των εγγράφων, αλλά δεν βλέπω αποτέλεσμα. Αν δείτε την παραγωγή μελιού, εδώ αναγράφεται από ένα χρόνο μέχρι απεριόριστο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να ε, περιπλέξει την ε, κατάσταση. Eh, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρεθήκανε ε, και βρέθηκε και απολυθωμένο μέλη σε διάφορες ε, αρχαιολογικές εξερευνήσεις που γίναν. Ποια είναι η ημερομηνία παραγωγής τότε που παράγεται το μέλι, δηλαδή η de facto παραγωγή ή το, το κουτί που πάει στο ράφι, γιατί μπορεί να διαφέρουν οι δύο ημερομηνίε κατά ένα χρόνο. Υπάρχουν επίσης ε, ε, παραγωγοί οι οποίοι ε, κάνουν προσμίξεις μελιού από τη δική τους χώρα και από μια άλλη χώρα και λένε ότι παράγεται από τη δική τους χώρα. Θα μπορείτε να μου πείτε τι συνέβη με το μέλι λοιπόν. Να, so ein naturverbundener Mensch wie der Alois Peter. Ε, Ένα άνθρωπο που δεσμευμένο με τη φύση, ο Alois Peter, έχει κάποιε ειδικέ ε, ε, ειδικά ενδιαφέροντα. Το μέλι από τη Σλοβενία θα μπορεί να το φάμε και μετά από 2.000 χρόνια. Δεν ξέρω τώρα αν το μέλι αυτό τον Φαραώ μπορούμε να το φάμε εμεί σήμερα. Ενδιαφέρον. Έχουμε και τον ε, διευθυντή κύριο Βούλινγκ από την Κομισιόν και μετά η κυρία Σόμερ να απαντήσει για το μέλι. Και κύριε Πίνε, έχω και εγώ μια ερώτηση. Αναφέρθηκε Φλιστάκης το θέμα των κεφαλαίων 6 και 7. Οι εθνικές ε, διατάξεις που θα επιτραπούν, τι γίνεται με το θέμα της αναμόνησης ε, δηλαδή εναρμόνιση με κοινοτικέ διατάξει και μετά έχουμε στο τυρί τη Σβίτσερη τρύπε τρύπε παντού γιατί υπάρχουν και εθνικέ. Πώ το βλέπετε. Oui, Monsieur le Να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε το λόγο. Άκουσα όλες τις ε, προτάσεις που υποβλήθηκαν με τις διάφορες προτάσεις συμβιβασμού. Νομίζω ότι δεν είχαμε δει τέτοια ε, σωρία τροπολογιών μέχρι τώρα, αλλά... Θα ήθελα για ε, να σας μιλήσω για την σήμανση. Μπροστά στο κάθε πακέτο, που αναγράφεται σε κάθε πακέτο. Νομίζω ότι θα πρέπει να ευχαριστούμε κυρία Ζόμερ και τα άλλα μέλη του Κοινοβουλίου που θεώρησαν ότι είναι σκόπιμο να υπάρχει μπροστά ε, η σύνθεση και τα συστατικά και λοιπά και όλα στην προστινή πλευρά δηλαδή του πακέτου. Γνωρίζετε ότι η θέση της Επιτροπής ε, ή μάλλον η Επιτροπή πάντα τάχθηκε υπέρ αυτών των εθνικών προγραμμάτων θεωρεί, θεωρώντας ότι θα πρέπει να φτάσουμε στην πλήρη εναρμόνιση. Μας φάνηκε δύσκολο στη μελέτη αντικτύπου να επιβάλλουμε ένα κοινοτικό πλαίσιο. Γι' αυτό λάβαμε υπόψη τα εθνικά προγράμματα με βάση την αρχή της ε, επικουρικότητας. Μετά από χρόνια όμως είδαμε να ανακύπτουν ε, διάφορα επιμέρους προγράμματα έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα κοινοτικό. Όμως αυτά τα εθνικά προγράμματα ε, ίσως προς το παρόν επαρκούν. Ως προς την επιλεξιμότητα έγινε μεγάλη συζήτηση στην Κομισιόν, Συμβούλιο κλπ. Θεωρούμε ότι το θέμα της αναγνωσιμότητας είναι μεγάλη σημασία. Γι' αυτό θα θέλαμε να λάβουμε υπόψη το μέγεθος των γραμμάτων. Το Συμβούλιο έχει υποβάλει μία πρόταση για το μέγεθος ε, των γραμμάτων. για να ξέρουμε τι θα γίνει όταν θα τυπωθούν οι ετικέτες. Θα ήθελα να σας πω ότι για μας είναι πιο σημαντικό να ξέρουμε ότι η προέλευση, τα στοιχεία προέλευσης δεν πρέπει να ε, παραπλανούν τον καταναλωτή, αλλά αναμένουμε τη δική σας ψηφοφορία καθώς και τη ψηφοφορία την τελική του Κοινοβουλίου, διότι η σήμανση προέλευσης θα πρέπει να μας απασχολήσει και μέσα στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, γιατί θα συντάξουμε μια πράσινη βίβλο και αναμένουμε με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις. Ως προς τις ε, απάτες, τις απομιμήσεις ε, προϊόντων και τροφίμων, θεωρούμε ότι έχουμε επαρκές ε, νομικό οπλοστάσιο, έτσι ώστε αν εφαρμοστεί σωστά από τις εθνικές ελεγκτικές αρχές, να, να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτά τα προϊόντα που παραπλανούν τον καταναλωτή έτσι ώστε να τηρεί το οποίο προέρχεται από, από, ουσίες, από φυτικές ουσίες να θεωρείται τυρί, ενώ στην ουσία δεν είναι. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε τους γενικούς ε, κανόνες έτσι ώστε να μην ε, εξαπατάται ο καταναλωτής σε σχέση με την νομοθεσία τροφίμων και θεωρούμε ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει να καταπολεμήσουν αυτές τις απομιμήσεις ε, τροφίμων έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η εξαπάτηση. Για το μέλι θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η νομοθεσία δεν επιβάλλει ε, μία προθεσμία κατανάλωσης. Ο παραγωγός ορίζει την προθεσμία κατανάλωσης του προϊόντος. Γίνεται υπό την δική του ευθύνη. Μετά από μελέτες για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος του κάθε είδους. Κάθε... Ε, αυτό ισχύει για τους ε, μελισσοπαραγωγούς, αλλά μπορεί να ισχύει για το γιαούρτι, για το κρέας, για το χοιρινό. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να γίνονται μελέτες για τον κύκλο ζωής του προϊόντος. 4, 5, 6 χρόνια, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μιλήσουμε για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν όμως κανόνες που ορίζουν το χρόνο ζωής και στην περίπτωση του μελιού ο παραγωγός θα πρέπει να ορίσει μία προθεσμία. Προθεσμία κατανάλωσης και θα πρέπει να αναγράφεται. Σε σχέση με την ε, οριζόντια σήμανση για τις εθνικές διατάξεις δηλαδή, υπάρχουν ε, διαδικασίες, προβλεπόμενες διαδικασίες με αυστηρές προδιαγραφές που σχετίζονται με θέματα υγείας του καταναλωτή, αλλά ακόμα και αν διαγράψουμε αυτό το κεφάλαιο, τα κράτη-μέλη μπορούν να ακολουθήσουν μια διαφορετική διαδικασία. Έχουμε την οδηγία 9834 για τις ρυθμιστικές προδιαγραφές τεχνικές προδιαγραφές και είναι μεγάλο πλεονέκτημα το ότι έχουμε αυτή τη διαδικασία, διότι μπορεί να γίνει διαβούλευση όχι μόνο σε επίπεδο επιτροπής, αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Θα παρακολουθήσουμε προσεκτικά την ψηφοφορία, τη δική σας ψηφοφορία αύριο, γιατί η κυρία Ζόμερ και ε, εσείς εμπλέκεστε ιδιαίτερα όσον αφορά αυτό το κείμενο. Αλλά όπως είπε και ο Επίτροπος Ντάλι, κατά την ακρόασή του, θα θέλαμε αυτή η νομοθεσία, αν εγκριθεί, να επιτρέψει στον καταναλωτή να έχει τις ε, περισσότερες δυνατές πληροφορίες για τα προϊόντα που έχει μπροστά του και ενδεχομένως αγοράσει. Δεν χρειάζεται όλες τις πληροφορίες, αλλά με βάση τα 500 εκατομμύρια καταναλωτών που έχουμε, που έχουμε να καλύψουμε, να ικανοποιήσουμε, θα πρέπει, θα πρέπει τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να καλύπτουμε τις ανάγκες τους. Μιλήσατε και για διατροφική αξία αυτό σχετίζεται και με θέματα επισήμανσης ή σήμανσης σε σχέση δηλαδή με τα συστατικά και τη διατροφική αξία. Δεν θα θέλαμε να παραπλονηθεί ο καταναλωτής από τις πληροφορίες αυτές. Θέλουμε μία ειλικρινή και πλήρη πληροφόρηση του καταναλωτή που να μην τον οδηγεί σε παραπλάνηση με βάση απατηλά στοιχεία που μπορεί να, προβάλλει, που να προβάλλουν οι παραγωγοί ή που, που παράλληλα μπορεί να κρύψουν και κάτι άλλο σε σχέση με το ε, προϊόν. Και αυτό αφορά ιδιαίτερα την ε, διατροφική αξία των προϊόντων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκαθαρίσαμε και το θέμα του μελιού. Νομίζω ότι ακούσαμε ό,τι είχαμε να ακούσουμε για σήμερα. Κυρία Ζόμερ, νομίζω ότι υπόθηκαν τα πιο σημαντικά στοιχεία. Θέλετε και πάλι το λόγο, ναι. Ναι, θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένα σχόλια. Αγαπητέ συναδελφέ Βέλμουτ, η σήμανση για τα φανάρια, η σήμανση φανάρια θα είναι μόνο για τα παρασκευασμένα προϊόντα. τα μεταποιημένα προϊόντα. Πού ξεκινάει η μεταποίηση όμως και πού σταματάει. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η σήμανση φωτεινού σηματοδότη για τα τρόφιμα. Το ξέρετε. Και γι' αυτό άλλωστε δεν εισήχθη και γενικά καθολικά στη Μεγάλη Βρετανία. Ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. Γίνεται μια συζήτηση στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά πολύ περιορισμένα και πιο περιορισμένα ακόμα στη Γερμανία και πουθενά άλλου. Και να πω και κάτι άλλο Πάντα με κατηγορείτε και πολλούς άλλους συνοδέλφους ότι ε, πάντα εισακούμε τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Το άκουσα και σήμερα πάλι. Να σας πω όμως το εξής. Αν υποστηρίζετε τις συνιστόμενες ε, ημιρήσεις ποσότητες, εσείς είσαστε που στηρίζετε τη μεγάλη βιομηχανία, γιατί οι μεγάλες εταιρείες ε, κατήρτισαν τον τις ημερήσεις συνιστόμενες ποσότητες. Το 20% απαρτίζουν αυτές οι, αυτές οι επιχειρήσεις. Ξεχνάτε όμως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απαρτίζουν το μεγαλύτερο σύνολο και αυτούς ακριβώς καταστρέφεται, θέσεις εργασίες καταστρέφεται με το GDA αυτό. Να το σκεφτείτε λοιπόν λίγο καλύτερα, σας προτείνω. Και δεν είναι εκατοντάδες αγαπητέ Πέτερ Λίζε, δεν είναι εκατοντάδες αυτές οι μικρές επιχειρήσεις, είναι χιλιάδες. Αυτός είναι ο κλάδος των τροφίμων. Και εκεί παράγονται οι περιφερειακές, οι τοπικές μας, ε, τα τοπικά μας προϊόντα. Δεν είναι μόνο πάντα η μεγάλη βιομηχανία, οι μεγάλες ε, επιχειρήσεις για την κρίστα κλάς και για την ε, επεξεργασία των επιφανειών. Υπάρχει σχετική... Υπάρχουν πάρα πολλοί αυστηρά, ε, όρια. Και νομίζω ότι αν και αυτό προσπαθήσουμε να το βάλουμε στην ετικέτα, θα προκαλέσουμε σύγχυση στον καταναλωτή. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο. Για την επισήμανση προέλευση, λέει ο συνάδελφο Νέλχερτ, ε, προάγει τον προστατευτισμό στα κράτη-μέλη για όλα τα προϊόντα. Ναι, αλλά, αλλά θεωρώ ότι το επίπεδο της πληροφόρησης του καταναλωτή και του προστατευτισμού αφετέρου είναι πολύ μικρή, αν θέλετε, η διαφορά σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, προέλευσης. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα χρειαστούμε μια μελέτη αντικτύπου. Αυτό αποτελεί μια ρεαλιστική ε, προσέγγιση. Για τις θρησκευτικέ ε, σφαγές τώρα. Καταρχάς η έκθεση αυτή αναβλήθηκε για την τρέχουσα αναβατική περίοδο και συμπεριέλαβα μια τέτοια προηγούμενη τροπολογία όπου αναφέρεται ότι το κρέας θα πρέπει να φέρει εκεί επισήμανση αν προέρχεται από ζώο που έχει σφαχτεί χωρίς με αμυστητοποίηση. Ε, και ξέρω ότι για παράδειγμα οι Ορθόδοξοι ε, Εβραίοι πρέπει να σφάζουν τα ζώα χωρίς αναισθησία, Ιδάλως το κρέας δεν είναι κοσέρ. Και τελικά εισάγονται τμήματα του κρέατος ε, τα οποία δεν μπορούν να φάνε οι Ορθόδοξοι Εβραίοι. Και ότι και γι' αυτό λοιπόν με τη δικασία αυτή ακριβένει υπερβολικά το κρέας κοσέρ για τους Ορθόδοξους Εβραίους. Αυτό να το σκεφτούμε ως θέματα. Για λόγους προστασίας των ζώων είμαι κατά της φαγής ε, χωρίς αναισθησία, πέρα από το θέμα των Ορθόδοξων Εβραίων. Δεν αναφέρομαι σε αυτό συγκεκριμένα, ανέφεραν συγκεκριμένο παράδειγμα κάποιος που ακολουθεί τα αρθόδοξα αυτά έθιμα μου είπανε ότι θα πρέπει να ακολουθεί οκτωετή εκπαίδευση προτού έχει δικαίωμα σφαγής. Αυτά λοιπόν τα έχουμε όλο υπόψη όταν θα ψηφίσουμε αύριο την 177 για το αλκοόλ, για το πνευμά. Θα θέλα να είμαστε συνεπείς και να εξαιρεθούν όλα τα αλκοολούχα προϊόντα και πάντα τίθεται το θέμα των αλκοπόψ. Αλλά συνάδελφοι, το γεγονός ότι περιέχεται ενόπνευμα, ούτως ή άλλως πρέπει να αναφέρεται στην επισήμανση. Μπορούμε να βάλουμε, αν θέλετε, και τις θερμητικές ε, τιμές, αξίες και τις θερμητικές αξίες, αλλά μήπως ε, δεν είμαι σίγουρη αν αυτό οφείλεται για το θέμα που αναφέρεται για το πρόβλημα των ε, νέων της νεολίας. Θα ήθελα να το εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε κατά πόσον ε, θα είχε νόημα να υπάρξει ανάλογη επισήμανση στα αλκοολούχα όπως και στα υπόλοιπα τρόφιμα. Για την επισήμανση των τροφίμων, ναι, το είχα πει και στην προηγούμενη των ε, απομιμήσεων. Το είχα πει ότι και το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει τι αγοράζει. Το θέμα δεν είναι να τα διώξουμε από την αγορά, το θέμα είναι να διευκρινίσουμε στον καταναλωτή ότι πρόκειται για απομίμηση, όχι για το γνήσιο προϊόν και μετά μπορεί να αποφασίζει ο καταναλωτής ανάλογα και με το πορτοφόλι του. Και κάτι άλλο για το μέγεθος ε, και την αναγνωσιμότητα. Είπατε ότι δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Φυσικά και μπορούμε να το αποφύγουμε. Αυτό το έχουμε κάνει άλλωστε έως τώρα. Και γι' αυτό και το αναφέρουμε και στις ενοποιημένε τροπολογίες ότι φυσικά το μέγεθος της γραμματοσυράς αποτελεί μόνο ένα στοιχείο της όλης αναγνωσιμότητας και υπάρχουν πάρα πολλά περαιτέρω στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λεφθούν υπόψη. Για το μέλι, για να μην συμπεριληφθεί στην ρύθμιση για την ε, ε, ημερομηνία λήξης. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να κοιτάξει και το Υπουργικό Συμβούλιο. Ξέρω ότι έχει μεγάλη ημερομηνία λήξη το μέλη και δεν ξέρω αν όντω πρέπει να επαφίεται στον παραγωγό αυτό, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως σε κάποιο άλλο επίπεδο θα πρέπει να περάσει μια πιο σαφή ρύθμιση. Και κάτι άλλο που ξέχασα να πω στην αρχή και με αυτό κλείνω. Υπάρχουν τροπολογίες για την επισήμανση προϊόντων με γενετικά τροποποιημένα συστατικά ζωικά προϊόντα όπου για παράδειγμα έχει τραφεί το ζώο με γενετικό τροποποιημένους οργανισμούς. Θεωρώ ότι αυτό είναι απαράδεκτο, δεν πρέπει να περιλαμβάνεται εδώ πέρα στο παρόν σχέδιο. Υπάρχει σχετικό νομοθέτημα για την ανιχνωσιμότητα και την επισήμανση των τροποποιημένων, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Δεν μπορούμε να περάσουμε τις διατάξεις μέσω του νομοθετήματος αυτού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, για τους επένους και περιμένω ε, αναμένω και τις υπόλοιπες ε, αμφισβητήσεις από τους υπόλοιπους και μην ξεχνάτε ότι και εγώ πολλά πράγματα έχω αναγκαστεί να ακούσω τα οποία δύσκολα μπορώ να δεχτώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ζωμάρ. Ε, με εδώ τη συζήτηση. Απόψε, αύριο θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Παρακαλώ όλοι να φέρετε τις κάρτες σας για την ψηφοφορία. Στις 9. Θα ξεκινήσουμε στην ώρα μας. Αύριο το ξαναλέμε. Πέρα συνεδρία.